Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει και είναι χρόνος και στιγμή κατάλληλη να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να κάνω πολλέ εισαγωγικέ παρατηρήσει για να γλιτώσουμε χρόνο και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στου πολλού εμπειρογνώμονε που έχουμε προσκαλέσει και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μα σωστά και έξυπνα. Η συγγήτρια είναι η Αγγέλικα Νίμπλερ από την Επιτροπή μα. Υπάρχει και η συντάκτρια της νομοδότησης, ε, κυρία ε, Ρίτα Κόρολα, φίλη της Επιτροπής μας. Και έχουμε και πολλούς εμπειρογνώμονες. Πρώτος εμπειρογνώμονα ο κύριος Μούρικ από την Τελεφώνικα. Αλλά θα δώσω καταρχήν το λόγο στην Αγγέλικα Νίβλερ να κάνει την εισαγωγή. denn den Termin hier den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten, für die äh, vereinzelten για τους ε, συναδέλφους ε, που είναι παρόντε, θέλω να πω ότι αύριο στι 12 είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ξέρω ότι είναι πολύ βραχυπρόθεσμο. Τώρα το ανακοίνωσα και δίνω το λόγο στην Αγγέλικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στην ακρόασή μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καταφέραμε να βολέψουμε την ακρόαση αυτή στο πρόγραμμά μας. Θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για την περιαγωγή που αποτελεί και βάση για την ακρόασή μας και θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Χαίρομαι που έχουμε πολλούς ε, παρευρισκόμενους γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Ε, σχεδόν 90% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν κινητό τηλέφωνο και ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο εξωτερικό αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με μία μελέτη του Ευρωβαρομέτρου, το, τα δύο τρίτα των καταναλωτών χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο σε περιαγωγή όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Και υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί οι οποίοι ε, κλείνουν το κινητό τους όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, ιδίως για την περιαγωγή δεδομένων, διότι οι καταναλωτές φοβούνται το σοκ του λογαριασμού που θα λάβουν όταν επιστρέψουν στη χώρα τους. Όταν επιστρέψετε στη χώρα σας μετά από την παραμονή σας στο εξωτερικό, δεν θέλετε να τρομάξετε από ένα τεράστιο λογαριασμό λόγω των τελών περιαγωγής. Στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά, στην ενιαία μας αγορά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιο κόστος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό για την ενιαία αγορά και για τους πολίτες. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν αυτό να το βελτιώσουμε. Το θέμα της περιαγωγή δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη το 2007 είχαμε τον πρώτο κανονισμό για την περιαγωγή και μετά δύο χρόνια αργότερα τροποποιήθηκε ο κανονισμός ε, και εκεί είχε προβλεφθεί ένα ανώτατο όριο και για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων SMS και για τις υπηρεσίες δεδομένων. Ε, τέθηκε ένα ανώτατο όριο χονδρικής αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανώτατο όριο λιανικής ε, για την περιαγωγή δεδομένων. Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια και τώρα ε, ξέρετε ότι όταν περνάτε τα σύνορα υπάρχει μήνυμα από τον πάροχο ε, που σας ειδοποιεί για το κόστος περιαγωγής στο εξωτερικό. Πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2011, η Επιτροπή ε, κατέθεσε την ενδιάμεση έκθεση για την κατάσταση των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα ναι, και οι πάροχοι κινητής ε, τηλεφωνίας θα πρέπει να προσαρμόσουν ε, ε, τις τιμές τους. Ήδη διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί οι τιμές περιαγωγής, αλλά υπάρχει ακόμη πεδίο βελτίωσης του ανταγωνισμού και οι τιμές ε, κινούνται κοντά στα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί. Δεν έχουν μειωθεί λοιπόν επαρκώς οι τιμές. Και με τη νέα πρόταση κανονισμού περιαγωγής ακριβώς αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή στην πρότασή της προτείνει μία διτή προσέγγιση να διατηρήσουμε τα ανώτατα όρια τα οποία υπάρχουν από πριν και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τον ανταγωνισμό στην αγορά με διαρθρωτικά μέτρα και συμπληρώνεται λοιπόν ο κανονισμός που υπήρχε για το ανώτατο όριο. Θεωρώ ότι όντως είναι σκόπιμο να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός στην αγορά κινητής τηλεφωνίας και σήμερα στη συζήτησή μας κατά την ακρόαση ακριβώς αυτό θα συζητήσουμε για νέους παρόχους στην αγορά περιαγωγής, για τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν για να προσελκύσουμε περισσότερους στην αγορά. Περνώ στα διαφορετικά μέτρα, τα μέτρα τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρετίζουμε και τα δύο αυτά διαφορετικά μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι η πρόσβαση στην περιαγωγή χονδρικής. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν πρόσβαση σε εναλλακτικούς παρόχους που δεν έχουν δίκτυο, που ονομάζονται εικονικοί πάροχοι για να μπορούν να μπουν στην αγορά της ε, περιαγωγής. Και στην έκθεσή μου υποστηρίζω ε, αυτή την προσέγγιση και τονίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια ρήτρα μη διακριτικής μεταχείρισης θα πρέπει να την χάνει ίσης μεταχείρισης λοιπόν και αυτός ο νέος πάροχος. Δεν είναι καινούριο στην οδηγία για την πρόσβαση ήδη από το 2009 όταν συμφωνήθηκε το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες υπήρχε και εκεί πάλι μια σχετική ρήτρα. Και εδώ νομίζω στο νέο κανονισμό για την περιαγωγή και πάλι πρέπει να βάλουμε κάτι αντίστοιχο. Το δεύτερο διαρθρωτικό μέτρο το οποίο προτείνει η Επιτροπή και το οποίο χαιρετίζω και εγώ στην έκθεσή μου είναι η, ο διαχωρισμός, είναι η αποδεσμοποίηση, το unbundling ο διαχωρισμό των υπηρεσιών περιαγωγή από τις υπόλοιπε υπηρεσίες. Δηλαδή ένας μεμονωμένος πελάτης θα μπορεί στην επικράτεια ενό άλλου κράτους μέλους ε, να συνάψει μία σύμβαση roaming με κάποιο πάροχο περιαγωγή στην άλλη χώρα. Κάποιο πάροχο δηλαδή που δεν θα είναι ο πάροχο τον οποίο έχει για την κινητή τηλεφωνία στη χώρα του. Η Επιτροπή στην έκθεσή της προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την αποδεσμοποίηση για το πώς θα μπορεί να γίνει και με, από τεχνικής πλευράς. Θα ακούσουμε πολλά περισσότερα και στην ακρόασή μας σήμερα. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για να είστε ενήμεροι. Ε, υπάρχει η, λύση των δύο ε, η των δύο ε, ταυτοτήτων, διεθνών ταυτοτήτων κινητού συνδρομητού ή της μίας ε, ταυτότητας, της ενιαίας ταυτότητας, Αυτά είναι θέματα που πρέπει να διαμορφώσει πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εθνικούς φορείς και με τον Μπέρεκ ε, και να ασχοληθούμε εμείς περισσότερο με την νομοθεσία. Να αφήσουμε τα θέματα του πώς θα γίνει στην πράξη στους τεχνικούς που έχουν την ε, τεχνογνωσία. Εμείς βέβαια είμαστε περίεργοι για το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και τι θα διαμορφωθεί τελικά. Και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας σήμερα στην ακρόαση σίγουρα θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Το επόμενο θέμα είναι το ανάτοτο όριο τιμών. θέλουμε ε, ακόμη πιο φιλόδοξες προτάσεις από ότι οι προτάσεις της Επιτροπής. Ο στόχος είναι μέχρι το 2015 το αργότερο να διαμορφωθεί μια κατάσταση κατά την οποία οι εθνικές τιμές, τα εθνικά τιμολόγια θα είναι παρόμοια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα χρειαζόμαστε πλέον τιμές περιαγωγής, θα έχουμε ίδιες τιμές σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση μέχρι το 2015 και για να το επιτύχουμε θα πρέπει τα σταδιακά βήματα που θα κάνουμε να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο θέλουν και οι οργανώσεις καταναλωτών. Ξέρω ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν την ίδια άποψη με τους καταναλωτές επί του θέματος, αλλά θα το δούμε και στην ακρόαση αυτό το θέμα. Θέλουμε να δημιουργηθούν κίνητρα για νέους παρόχους στην αγορά περιαγωγής, για να μπορούν να μπουν και νέοι πάροχοι, να δούμε ποια θα είναι η σχέση μεταξύ των τιμών χονδρικής και των τιμών λιανικής. Ίσως να έχει ο πρόεδρος ε, εδώ δίπλα μου διαφορετικές προτάσεις από μένα, αλλά γι' αυτό θα κάνουμε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, γιατί μπορεί να έχουμε διεστάμενες απόψεις. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί θα θέλει να μιλήσει και η συνάδελφος η κυρία Κορόλα. Το επόμενο σημείο που θα αναφέρω πολύ σύντομα είναι η διαφάνεια. Θέλουμε να έχουμε διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών. Πολλά θέματα τα οποία συζητάμε στην Επιτροπή μας συζητάμε και η κυρία Κόρολα στο πλαίσιο διαφορετικής έκθεσης, όχι μόνο ε, για να αποφύγουμε αυτό το σοκ που προέρχεται από το λογαριασμό ε, από τέλη περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη χρήση κινητού σε άλλες χώρες, ε, στις χώρες της Βορειοαφρικής, και σε άλλες χώρες τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι η τιμή είναι 50 cents. Είναι, συγγνώμη, τώρα υπάρχει ένας περιορισμός 50 ευρώ ε, για να προστατεύεται ο καταναλωτής και να μην υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση από 50 ευρώ, επομένως να μην ξαφνιάζεται από πολύ ψηλό λογαριασμό όταν επανέρχεται στη χώρα του. Αλλά και αυτό ακόμη θα μπορούσε να ρυθμιστεί και θα μπορούσαμε να έχουμε και κάτι καλύτερο προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ ως γενική παρουσίαση της έκθεσης. Και εγώ έχω τρία ερωτήματα τα οποία με απασχολούν και θα ήθελα να συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες. Το θέμα του πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά, στον τομέα των αερομεταφορέων, παραδείγματο χάρη. Δείτε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Πριν από 10 χρόνια δεν θα είχε φανταστεί κανείς ότι από το μόναχο στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να κοστίζει 20-30 ευρώ το ταξίδι με αεροπλάνο και το άνοιγμα της αγοράς ε, με τις φτηνές ε, αεροπορικές εταιρείες ε, έχει δώσει ένα νέο άνοιγμα στην αγορά. Έχουν διπλασιαστεί οι πάροχοι υπηρεσιών. Θα ήθελα να μπορούσαμε μια αντίστοιχη εξέλιξη να έχουμε και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω την άποψη όλων των συμμετεχόντων στο πάνελ. Πώς σας φαίνεται μια τέτοια πρόταση. Επίσης το θέμα των ε, τεχνικών προδιαγραφών είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει η Επιτροπή μαζί με τον ε, Ευρωπαϊκό Φορέα, τον Μπέρεκ, ε, να συζητήσουν αυτά τα θέματα και το θέμα των ανωτάτων ορίων τιμών είναι το επόμενο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Ο συνάδελφο Ρούμπιχ την προηγούμενη φορά μα είχε δώσει κάποιες τιμέ ε, και από την Αγγλία. Εσεί, κύριε Ρούμπιχ στην Αυστρία αλλά και εγώ στην Γερμανία ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ προσφορέ ε, για το εγχώριο κοινό. Υπάρχει προσφέρουν τιμές 8,80 ευρώ το μήνα για ένα έξυπνο κινητό που περιλαμβάνει 1000 λεπτά κλήσεων, 1000 μηνύματα SMS και 1000 MB στην τιμή των 8,80 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν κάποιες καταποκοπή τιμές για τους επιχειρηματίες που παρέχουν ευνοϊκά προτερήματα και στο εξωτερικό όταν κανείς κινείται από την άλλη μεριά των συνόρων ε, υπάρχουν τιμές για υπάρχουν διαφορετικές τιμές ε, από την άλλη μεριά των συνόρων και μπορεί, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσο φτηνές τιμές μέσα στην ίδια χώρα, να πληρώνω το διπλάσιο ή τριπλάσιο για λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε παραδεκτό στην ε, ενιαία αγορά. Μέχρι τώρα δεν ε, τα έχουμε διευκρινίσει και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στη σημερινή ακρόαση. Εγώ μπορώ να μείνω μέχρι τις 5 γιατί έχω πτήσει αργότερα και πρέπει να πάω στο Μόναχο, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγέλη Νίμπλα, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε στην ακρόαση και πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Μούρικα από την Τελεφώνικα. Θα σας παρακαλέσω να τηρήσετε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Να παρευρεθώ εδώ. Όταν ε, μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια από την ε, εκ μέρους τους τηλεφώνικα, σκέφτηκα τι εννοούμε με το roaming 3, 3, με την περιεγωγή 3, γιατί φαίνεται σαν να είναι μια από αυτές τις ε, ταινίες sequel του Hollywood ε, και η περιαγωγή 3 είναι πραγματική ευκαιρία. Η κυρία Κρούς ε, παρουσίασε μια πρόταση που διαφέρει από τις προηγούμενες και προσπαθεί να εξεύρει μια διαρθρωτική λύση. Έτσι λοιπόν, ε, για να τελειώσει το ετήσιο καθορισμός τιμών που έχουμε τώρα, προσπαθεί δηλαδή να βρει μία μόνιμη λύση. Ήμασταν κάπως σκεπτικοί στην αρχή, αλλά μετά από πολλή ανάλυση και σκέψη πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η διαφορετική λύση. Είμαστε λοιπόν αρκετά θετικοί απέναντι στην πρόταση Κομισιόν και την υποστηρίζουμε ευρέω. Βέβαια πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες, αλλά γενικά την υποστηρίζουμε. Και ένα από τα κύρια μηνύματα που θα ήθελα να ζητήσω από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να δείτε αυτή την πρόταση με έναν ε, ολιστικό τρόπο. Δηλαδή, να τη δείτε στο σύνολό τη, ε, όχι να τη δείτε ε, στα επιμέρου σημεία τη ένα προ ένα. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει η διαρθρωτική λύση και θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα συνεισφέρουν στο να λύσουμε το πρόβλημα της περιαγωγή. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πιστεύουμε ότι μπορούμε να βάλουμε στο μείγμα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ένα είναι κάτι που θα αναφέρω και κάπως αργότερα νομίζω ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει μία εξαίρεση για τους πάροχους που ε, χρεώνουν ε, τιμές ε, κοντά στις εγχώριες τιμές. Έτσι λοιπόν αυτό θα ήθελα να το αναφέρω. Και δεύτερον, Ακούω πάρα πολλά και ψηλέ ε, τιμέ για τα δεδομένα και αυτό ισχύει. Αλλά αυτό που είδαμε επίση τα τελευταία χρόνια είναι ότι πολύ γρήγορα πέφτουν οι τιμές για τα δεδομένα τελευταία. Έτσι λοιπόν ε, είδαμε ναι, γίνονται νέες προσπάθειες στην αγορά για να ε, τεθούν σε εφαρμογή νέα σχέδια τιμών για την περιεγωγή δεδομένων και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αυτές οι τιμές μειώνονται και εμείς ε, ως τηλεφωνικά μέχρι το 2015 πιστεύουμε ότι η αγορά θα παράσχει περιεγωγή των δεδομένων με τιμές που θα είναι πάνω κάτω ίδιες όπως ε, και οι τιμές σε εσωτερικό επίπεδο. Τώρα, η ερώτηση που πρέπει να ρωτήσετε, πιστεύω, τους αυτούς σας, ε, ως ε, κοινοβούλιο είναι, πιστεύετε αν θα, θα λειτουργήσει η διορθωτική λύση ή όχι. Αν πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει η διορθωτική λύση, τότε η αγορά θα μειώσει, θα οδηγήσει στη μείωση των ε, τιμών λιανικής. Ε, η αγορά θα λειτουργεί και τότε δεν έχει σημασία τι ανώτατορια τιμών θα βάλετε στον κανονισμό. Και εμείς ε, έτσι το βλέπουμε, δεν έχει σημασία αν είναι 20, 25, 50 cents λεπτά, γιατί η αγορά θα καθορίσει τις τιμές και, αυτό θα είναι, και αυτές θα είναι κατώτερες από το όριο τιμών. Έτσι λοιπόν. Τώρα να θέσετε ανώτατο όριο ασφαλείας, γιατί θέλετε να δώσετε μία εγγύηση στους καταναλωτές, αλλά για μας η πρόταση της Κομισιόν ε, μας κάνει σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια τιμών. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα ανώτατα όρια τιμών που θέτετε ε, ευνοούν ε, νέους παίκτες να μπουν στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να θέσετε τέτοια όρια έτσι ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον περιθώριο για τους νέους ερχόμενους. Γιατί αν δεν έρθουν ε, νέοι ε, στην αγορά, δεν μπορείτε να έχετε την διαρθρωτική λύση. Δεν πιστεύουμε επίση ε, ότι μπορείτε να πείτε αν, ότι, αν δεν πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτή η διορθωτική λύση, τότε ε, μην την εκπονήσετε, γιατί είναι ακριβή ε, να εφαρμοστεί από τους παρόχους, κυρίως για τους μικρούς παρόχους. Βρείτε λοιπόν έναν ευφυή τρόπο να καθορίσετε τις τιμές, αλλά μην υιοθετήσετε τη διορθωτική λύση. Πρέπει να κάνετε μία επιλογή, νομίζω, λοιπόν, ως Κοινοβούλιο, γιατί αν θα έχετε μία διορθωτική λύση συν ανώτατο ρε τιμών που θα δίνει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά ή θα κάνετε ρύθμιση των τιμών. Και ειλικρινά, αν δούμε τις τελευταίες προτάσεις ε, που κυκλοφόρησαν, ε, ξέρω ότι δεν έχουν ε, ψηφιστεί, η εντύπωσή μου είναι ότι έχετε επιλέξει το τελευταίο, δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργήσει η διαφορετική λύση και ότι χρειάζεται ένα τεταρίο τιμών που να είναι υπερβολικά αυστηρά. Δείτε τον πίνακα εδώ, κυρίως ε, στα δεξιά. Εδώ το Κοινοβούλιο έχει επιλέξει στην περίπτωση αυτή ανώτατο ρυθμόν 10 cents ε, για ε, τις φωνητικές κλήσεις και αυτό είναι που είχε η Κομισιόν κατά νου αν δεν ε, είχε εισαγάγει μια διαφορετική λύση. Έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε για ξεκαθαριστημές. Και επίσης ζητήσαμε από μια ανεξαρτητή την A.T. Kearney, να εξετάσει το business case για έναν επαναπολιτή, για ένα MVO, για έναν εικονικό πάροχο. Και βλέπετε εδώ ότι οι περισσότεροι εικονικοί πάροχοι, εκτός από τους ε, πάρα πολύ χαμηλού κόστους, δηλαδή εκεί όπου έχουμε πάρα πολύ μικρό προσωπικό δεν θα μπορέσουν ε, να έχουν κέρδος σε κανένα στάδιο. Έτσι λοιπόν από τα κυρία μηνύματα για μένα είναι να έχουμε λογικές, ε, λογικά όρια τιμών και να δίνεται στους παρόχους περιθώρια που να επιτρέπουν την είσοδο στην αγορά γιατί χωρίς αυτά τα περιθώρια δεν θα λειτουργήσει η διαφορετική λύση. Και νομίζω ότι είναι, αυτό είναι το κύριο. Ακόμη και αν θέσετε ε, πιο ψηλέ τιμέ, θα υπάρχει ανταγωνισμό ε, για την κατάργησή του και αν δεν ε, μειωθούν μέχρι το 2015, τότε μπορείτε να το ρυθμίσετε στην αναθεώρηση το 2016. Έτσι λοιπόν μπορείτε να έχετε την ευκαιρία νέα προσαρμογή. Και κάτι τελευταίο, πιστεύουμε ότι οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν και μια εναλλακτική η τιμή για την εφαρμογή διαθροτικής ε, λύσης, το τίμημα, είναι αρκετά μεγάλο. Δεν ε, είναι τόσο σημαντικό αυτό να έχετε 25 εκατομμύρια πελάτες, αλλά αν είστε πάροχος με 300.000 ε, πελάτες, τότε είναι σημαντικό αυτό το κόστος. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές οι ίδιοι πάροχοι, πιο μικροί, είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως σκέφτονται μπορούμε να μπούμε στην αγορά με ένα σχέδιο τιμών ε, και με ένα σχέδιο τιμών για την περιαγωγή, δηλαδή με το οποίο χρεώνουμε πάνω κάτω το ίδιο όπως για τα, στην εγχώρια περίπτωση. Κατά την άποψή μα, αυτό θα πρέπει να το κολοσυρίσετε. Συνάδει απόλυτα με το ψηφιακό θεματολόγιο τη Κομισιόν, τη κυρία Κρού, και κάτι τέτοιο θα έδινε όθηση ανταγωνισμού στην αγορά γιατί αυτοί οι μικροί πάροχοι θα είχαν ε, μια εναλλακτική να προσφέρουν ε, στην αγορά και πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή εναλλακτική να επιτρέψετε στους παρόχους να ρυθμίζουν ίδια τη μοίρα τους, για να το πούμε έτσι. Τώρα, συμπεράσματα. Πιστεύουμε καταρχήν ότι η διευθυντική λύση μπορεί να λειτουργήσει αν ε, σχεδιαστεί σωστά, αλλά χρειάζεται ενώ το τώρα δημόσιο που να αφήνει περιθώριο για την προσέλκυση επενδυτών. Και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι αυτά τα όρια τιμών δεν πρόκειται να ελκύσουν ως επενδυτές. Πρέπει να κάνετε μια επιλογή για το αν θα τολμήσετε να προχωρήσετε με ρύθμιση των τιμών όπως ε, είδατε ή θα επιλέξετε μια βιώσιμη και μόνιμη λύση, την οποία σκοπεύουμε εμείς, Νομίζω ότι πρέπει να εισαγάγουμε αυτή την εξαίρεση για αυτή την τιμολόγηση που είναι κοντά στις ε, χώριες τιμές και νομίζω ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά και το υποστηρίξουμε όλο αυτό το εγχείρημα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά και πιστεύω ότι καθυστέρησε ένα λεπτό. Λυπάμαι. Ε, Σας ευχαριστούμε. Μια πρόταση είναι ε, να αφήσουμε τους ομιλητές να λαμβάνουν το λόγο ο ένας με τον άλλον. So, Sorry. I'm just going to try to find you. Okay, the next is. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Εμμάνουελ Φόρεστ. Technik klappt? Nein. Angelika benutzt jetzt ja auch noch den Computer. I don't know. Perhaps first sit Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Φόρεστ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η Μπούγκ Τελεκόμ πάντοτε στήριζε το στόχο της Κομισιόν για μείωση των τιμών περιαγωγής προς όφελος των καταναλωτών. Στηρίζουμε πλήρως λοιπόν τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου. Φαντάζομαι ότι ο επόμενος ομιλητής ε, θα είναι πρόσωπος ε, της ε, εταιρείας Transatel. Πριν από κάποια χρόνια έχουμε, συνάψαμε και ένα συμβόλαιο με την εταιρεία αυτή για να υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές πάλι στον τομέα της περιαγωγής. Ο εξαφωνήμων συνάδελφος ε, θα σα τα πει αυτά αργότερα. Βλέπουμε ότι η διαθροπική λύση που προτείνει η Κομισιόν είναι πολύπλοκη, ιδιαίτερα πολύπλοκη και ουσιαστικά αποτελεί ένα πολύ ισχυρό, αν θέλετε, φάρμακο για το πρόβλημα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι η χοντρική πρόσβαση θα μπορούσε να έχει κάποιες ε, αρνητικές συνέπειες στην αγορά και... From my colleague of Telefonica to uh, achieve the goal of the digital agenda και θα πρέπει οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου να μπορέσουν να επιτευχθούν ταχύτερα και ευκολότερα. Θεωρούμε ότι η αρχή της αποσύνδεσης είναι πολύπλοκη, είναι πολύπλοκη λύση, πολύπλοκη για τους πελάτες, τη πλειονότητα αυτών που δεν θα καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν άλλη εταιρεία για τις εγχώριες υπηρεσίες και άλλη εταιρεία για τις διεθνείς. Θα είναι πολύπλοκο και για τους λιανοπολιτές να μπορέσουν να ε, θέσουν στο εμπόριο αυτές τις υπηρεσίες. Δέκα δις είναι οι νέες επενδύσεις για τα συστήματα και για την ασφάλεια, δηλαδή που θα χρειαστούν πολλά χρήματα και για τις επενδύσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι ζήσαμε στο παρελθόν την επιλογή παρόχων στη σταθερή τηλεφωνία. Δεν στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η πρόταση της Κομισιόν με την αρχή της αποσύνδεσης, της αποδεσμοποίησης είναι λίγο πολύ η ίδια. Άρα μπορεί να λειτουργήσει κακά, όσο κακά λειτουργήσει και για την σταθερή τηλεφωνία. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό επίσης, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, γιατί όπως είπα υπάρχει σημαντικό κόστος εφαρμογής και αυτό το κόστος εφαρμογής θα είναι αναλογικά υψηλότερο για μικρότερους ε, παρά για μεγαλύτερους παρόχους. Εξού και φοβούμε ότι οι μεγαλύτεροι πάροχοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες ε, ε, φαίνεται να δέχονται την πρόταση της Κομισιόν για αυτό το λόγο. Κάτι πολύ σημαντικό, το brand name, το εμπορικό, η εμπορική ονομασία κανείς δεν μπορεί να προφέρει το όνομα Bouygues. Γι' αυτό και η Bouygues Telecom δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε άλλη πάροχη. Θα ήταν ε, ίσως ε, πιο εύκολο να είχαμε ένα όνομα όπως Telefonica, Orange. Ε, τέλος πάντων δεν θέλω βέβαια να κάνω διεύθυνση στους ανταγωνιστές μου, αλλά τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά τώρα την χοντρική πρόσβαση και αυτή θα είναι και η εστίαση που θα έχει η ομιλία μου, στην πρώτη μου ε, πρόταση να σας δώσω ένα παράδειγμα. μπορεί να υπάρξουν ε, κάποιοι εναλλακτικοί πανευρωπαϊκοί πάροχοι για να παρέχουν ευρωπαϊκές υπηρεσίες παραγωγής στους καταναλωτές. Θα μπορούσαν να ανεβούν τέτοιοι πάροχοι, αλλά είναι θεωρητικό αυτό το ενδεχόμενο. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αγοράσουν μια κάρτα SIM από έναν πάροχο από το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα. Οπότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την πανευρωπαϊκή υπηρεσία όχι για την περιαγωγή αλλά και για την ε, εγχώρια ε, χρήση, για τα εγχώρια τηλεφωνήματα. Πώς θα μπορούσαμε νομικά λοιπόν να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ παραδείγματος ενός Ιρλανδού υπηκόου με την Πανευρωπαϊκή Υπηρεσία από Λουξεμβουργιανό πάροχο με περιαγωγή στη Γαλλία και πώς θα τον διακρίνουμε από ένα Γάλλο υπήκο κάτοικο Γαλλίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε μια κάρτα σήμα από το Λουξεμβούργο και παράνομα χρησιμοποιεί τις πανευρωπαϊκές αυτές υπηρεσίες ως εγχώριες υπηρεσίες. Φοβόμαστε λοιπόν ότι αυτή η χοντρική πρόσβαση τελικά δεν θα είναι πανευρωπαϊκή πρόσβαση, αγροτικές υπηρεσίε για το roaming, αλλά γενικά πανευρωπαϊκή πρόσβαση ε, σε χοντρική. Άρα θα πρέπει ε, πρώτα να δούμε τις, ε, τα, τις ιδέες μας, αλλά πρώτα να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την τη της Πρώτα απ' όλα είναι αντιφατικό με το γεγονός ότι η πρόσβαση στην αγορά εξαιρείται από τον κατάλογο των σχετικών αγορών από την Κομισιόν σε εθνικό επίπεδο για τους σκοπούς της ανάλυσης αγοράς. Δεύτερον, η αρχή της επικουρικότητας ε, δεν ε, ε, θα έπρεπε να τηρεί κανονικά οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες και επίσης πηγαίνει πολύ μακριά. Γιατί, γιατί όπως είπα έχετε αυτό το κόλπο. Δηλαδή το τέχνασμα, ο Γάλλος υπήκος να μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σήμα από το Λουξεμβούργο, όπως σας είπα, με την πανευρωπαϊκή υπηρεσία είτε από το Λουξεμβούργο είτε από την Ιρλανδία από ένα τέτοιο πάροχο, από πάροχο άλλης χώρας. Έγινε ανάλυση άγορας από την ε, Κομισιόν. Το Staff Working Paper της Κομισιόν του Ιουλίου δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, στη σελίδα 35, αν το έχετε διαβάσει θα δείτε ότι εξετάστηκαν τρεις λύσεις. Εγώ τις δύο τελευταίες διάβασα. Ή περιορισμένη χοδρική πρόσβαση για το roaming, είτε πρόσβαση για όλες τις κινητές υπηρεσίες. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή η οποία προκρίνεται από την Κομισιόν για την περιαγωγή δηλαδή. Γιατί η Κομισιόν όμως αρνείται την τρίτη λύση, γιατί την απορρίπτει μάλλον την τρίτη λύση για όλες δηλαδή τις υπηρεσίες, γιατί βρήκαν ένα μειονέκτημα. Αν δεν περιορίζεται αυτή η επιλογή στις υπηρεσίες ε, περιαγωγής, θα μπορούσε να στριβλώσει ή να καταστρέψει τον ανταγωνισμό στις εγχώριες αγορές και άρα θα υπερβεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό ε, την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το roaming. Επομένως, ε, η Κομισιόν τελικά δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν γνήσια πανευρωπαϊκή πάροχη και για την περιαγωγή αλλά και για τις εγχώρες υπηρεσίες. Το γράφει και η διαπιτροπή ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Αυτά λοιπόν τα βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Και να πω επίσης, κατακλείδη ότι για μας και πάλι δεν κάνω διαφήμιση, η καλύτερη πάροχη θα μπορούσε να είναι το Google ή η Apple. Γιατί είναι πολύ εύκολο να επιλέξει κανείς τις τιμές ε, για το roaming ε, με την εφαρμογή iTunes, για παράδειγμα. Οπότε Google και Apple είναι πολύ πιο εύκολο να μπουν ε, στην ευρωπαϊκή αγορά ως MVNOs εικονική πάροχη όχι όμως για την Πανευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιαγωγή, αλλά και για τις εγχώριες υπηρεσίες. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο από νομικής πλευράς να κάνει κάποιος τη διάκριση μεταξύ υπηρεσίας roaming και εθνικής υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το roaming data cap, ένα μήνυμα έχουμε να δώσουμε προς την ε, Κομισιόν και το λέμε εδώ και χρόνια. Θεωρούμε ότι με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 3G και 4G, δεν μιλάμε πλέον με megabyte ή gigabyte. Η... Κάτι που είναι πολύ δαπανηρό για έναν πάροχο είναι να κάνει roll out του δικτύου, να δώσει πρόσβαση στον πελάτη, όχι να παράσχει ένα megabyte, ένα gigabyte παραπάνω. Επομένως, για την χρέωση των δεδομένων roaming θα μπορούσαμε να, δούμε, να κάνουμε αυτό που κάνουν τα ξενοδοχεία. Να αγοράζει δηλαδή κάποιος ε, σύνδεση για ένα, μια ώρα, μια μέρα, ένα μήνα και δεν ξέρω εγώ πόσο. Θα μπορούσε αυτό να είναι δυνατό, αλλά μόνο εάν οι άνωτες ε, τιμές εξελίσσονταν προς ένα τέτοιο ε, σχήμα. Δηλαδή να υπάρχει μια σταθερή χρέωση πρόσβασης. Δηλαδή κάποιος να πληρώνει στον πάροχο το πάγιο είναι την ε, τιμή αναμονάδα, ένα δεδομένο μεγαμπάιτ για παράδειγμα. Αλλά με τον τρόπο αυτό νομίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει οι πάροχοι να έχουν τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμα να υιοθετήσουν τα πλέον κατάλληλα ε, σχήματα τιμολόγησης. Ολοκληρώνοντας να πω Βέβαια είναι πολύπλοκα όλα αυτά τα θέματα. Η δική μας ιδέα ήταν ε, ότι ο σωστός τρόπος Βέβαια είναι μια θελοντική πρόταση. Η Buick Telecom αλλά και άλλοι μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν αυτή την πρόταση. Να εφαρμόσουν το ψηφιακό θεματολόγιο το 2015. Η ιδέα μας λοιπόν ποια είναι. Ο πάροχος μπορεί να αποφασίσει ή ίσως και να εξαναγκαστεί να χρεώνει ένα ακόμη πάγιο ε, ποσό για την γεωγραφική επέκταση του σχήματος ε, των τιμών, είτε να είναι αποθεσμοποιημένο, είτε όχι. Εγώ σα έδωσα ένα παράδειγμα. Είμαι Γάλλο υπήκο, πηγαίνω στη Γερμανία, ταξιδεύω στην Ευρώπη τέλο πάντων. Άνε για μία μέρα, με ένα ευρώ. Μπορώ να έχω λοιπόν ε, την γεωγραφική επέκταση των υπηρεσιών. Άρα έχω μια, ένα γεωγραφικη επεκταση των υπηρεσιων αρα εχω ενα γνησιο ε, μια γνήσια χρέωση πανευρωπαϊκή. Αυτό χρησιμοποιήθηκε πριν από 10 χρόνια για να πάμε στη δημολόγηση για ένα ε, δευτερόλεπτο ή ένα λεπτό. Ένα οψιον φυ μας υποχρέωσαν οι αρχές να, ε, να βάλουμε και σιγά σιγά εξασλήφθηκε αυτή η χρέωση. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν, τηρώντα και το ψηφιακό θεματολόγιο, να υιοθετήσουμε πραγματικά τιμέ πανευρωπαϊκέ για όλο την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουν οι ομιλίτες στο πάνελ λοιπόν. Ζακ Μοντιφάη της Transatel. Έχετε το λόγο και τον υπολογιστή. Have you I do right now. Voilà. he had his, presentation. Yeah, that's my presentation. So that's so, okay, that's so Good afternoon. My name is Jacques. Καλησπέρα. Ζακ Μπονιφέ είναι το όνομά μου. Είμαι πρόεδρος μιας ένωσης εικονικών παρόχων στη και η της Τρανζατέλ. είμαι ως επιχειρηματίας. Σε έξι χώρες λειτουργούμε, 8,4 δις ευρώ είναι ο κύκλος εργασιών μας. Είναι μια πανευρωπαϊκή εταιρεία. Προσφέρουμε υπηρεσίες σε πολίτες που ταξιδεύουν συχνά και που περνάνε τα σύνορα συχνά. Αυτό που ήθελε να εφαρμόσει η Vivian Redding τα τελευταία χρόνια, το κάνουμε εμεί ε, γύρω στα 10 χρόνια τώρα και θα σα εξηγήσω λίγο περισσότερο τι κάνουμε. Είμαστε και εταιρεία enabler, δηλαδή ε, δίνουμε προϊόντα σε εικονικού παρόχους. Έχουμε 17 εικονικούς παρόχους στην Ευρώπη πολλούς συνδρομητές σε έξι διαφορετικές χώρες ε, και υποδομές που συνδέονται με 8 δίκτυα στην Ευρώπη βασιζόμαστε σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλής ταυτότητας χρήστη. Δηλαδή στην κάρτα SIM που βρίσκεται σε αυτό το κινητό μπορώ να έχω πέντε αριθμούς από πέντε διαφορετικές χώρες. Ένα γαλλικό, ένα βελγικό, ένα ολλανδικό, λουξεμβουργέζικο και ελβετικό. Buick, Bobby Star, Orange για την Ελβετία, Tango για το Λουξεμβούργο και Telford KPN για την Ολλανδία. Έχω και ελβετικό αριθμό, όπως σας είπα. Η Ελβετία δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί αυτή η λύση μας και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνουμε μία κάρτα SIM και μία συνδρομή στον τελικό χρήστη δίνουμε τη δυνατότητα για χρήση σε εθνικό επίπεδο και σε περιαγωγή και την επιλογή αυτή την κάναμε για οικονομικούς λόγους για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες οι υπηρεσίες μας και θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και στις ΗΠΑ Πολιτείες και στο Ισραήλ και να προσφέρω τοπικές τιμές στις ΗΠΑ Πολιτείες και στο Ισραήλ προς Ευρωπαίους πολίτες. Να έχω δηλαδή τοπικές τιμές. Δεν το κάνω γιατί προς το παρόν δεν έχουμε τόσο μεγάλη κάλυψη. σα είπα λοιπόν ότι απευθυνόμαστε σε διαμεθοριακό πληθυσμό για Γάλλους που δουλεύουν στην Ελβετία καθημερινά, για ε, πολίτες που κινούνται προς το Λουξεμβούργο. Δίνουμε εκπτώσεις 50% στην περιαγωγή και θα μπορούσαμε να δώσουμε και μεγαλύτερες αν είναι απαραίτητο. Ε, 95 ευρώ το μήνα είναι το ARPU, το μέσο έσοδο αναχρήστη και το περιθώριο κέρδους μας είναι περίπου 40%. Βλέπετε ότι μπορώ σε λιγότερο από 12 μήνες να μπορέσω να καλύψω το κόστος ε, κτήσης. Είναι οικονομικά δεδομένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να δούμε ποια είναι η σωστή τιμή για το ε, σωστό ανώτατο όριο για την περιαγωγή. Οι λύσεις που έχουμε δεν είναι λύσεις μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για εκτός ε, Ευρώπης. Θα σας πω γιατί η Τρανζατέλ δεν είναι μεγαλύτερη, γιατί έχουμε λιγότερους από 10.000 συνδρομητές. Ο λόγος είναι απλός. Προσπαθήσαμε πολλές φορές επί χρόνια να δουλέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν τα καταφέραμε, στη Γερμανία δεν τα καταφέραμε, στην Ισπανία δεν τα καταφέραμε, στην Ιταλία δεν τα καταφέραμε. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να περιοριστούμε μόνο στη Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και πρόσφατα στην Ελβετία. Εφτά χρόνια χρειάστηκα για να, κάνω, να βρω μια συμφωνία στην Ελβετία. Επίσης το ότι δεν μπορούσα να κάνω συμφωνίες περιαγωγής με χώρες όπως η Γερμανία γιατί θα μπορούσα να, να κάνω συμφωνίες περιαγωγής με κάποιο πάροχο στη Γερμανία και να μπορώ να προσφέρω καλύτερες τιμές στο Γάλλο ή στο Βέλγο πελάτη μου που πάει στη Γερμανία. Έχουμε λίγους συνδρομητές, λιγότερο από 10.000, ενώ η αγορά στόχους μου θα μπορούσε να είναι δυνητικά 3 εκατομμύρια πελάτες. Δεν είχα μεγάλη υποστήριξη από, τις, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτό πρέπει να το πω, παρότι συναντήθηκα με τη Vivian Redding. Και εγώ τι ζητούσα, δεν ζητούσα ρυθμιστική παρέμβαση, ζητούσα κάποιο είδους δημόσια δήλωση που θα έλεγε ότι ένας πανευρωπαϊκός εικονικός πάροχος με πολλαπλό IMSI θα ήταν μια καλή λύση. Και δεν είμαστε η μόνη εταιρεία εμείς η Transatel, ξέρω και άλλους και πολλοί που έχουν χρεοκοπήσει γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Είναι μια λύση εφικτή, αυτό το οποίο προσφέρει η Τρανζατέλ, αλλά χρειαζόμαστε κάποια υποστήριξη ώστε οι πάροχοι σε άλλες χώρες να θελήσουν να κάνουν συμφωνία μαζί μας. Θα πρέπει να ενθαρρύνετε λοιπόν τους παρόχους. Αν θα το κάνετε με κάποια ρύθμιση ή με κάποια δήλωση, δεν ξέρω, πάντως κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μου σε γενικές γραμμές και θα περάσω στις τρεις διαφορετικές λύσεις που προτείνονται. Προτείνονται τρεις λύσεις, πρέπει να σας πω. Όλες οι λύσεις που έχουμε ε, στην ε, Transatel είναι ε, καλές, έχουν δουλέψει τα τελευταία δέκα χρόνια, επομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα επιπλέον μοντέλο. Το τωρινό μοντέλο θεωρώ ότι είναι κάπως αδύναμο, γιατί είναι ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μα που υπάρχει τώρα. Για το local breakout πρέπει να πω ότι είναι κάπω επικίνδυνο όσον αφορά το τελικό χρήστη. Ποια είναι η καλύτερη εταιρεία που θα δώσει το καλύτερο προϊόν, η Apple και η Google με τα Android. Αν εφαρμόσουμε το local breakout, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για την Google και για την Apple. Δεν είμαι λοιπόν πολύ βέβαιος ότι θέλουμε ε, εμείς να μειώσουμε το έλλειμμα της Καλιφόρνιας και να δώσουμε λεφτά στην Google και στην Apple, γιατί αυτό θα συμβεί. για τους Αμερικάνους και για τους Κινέζους που έρχονται στην Ευρώπη θα είναι τέλεια γιατί θα υποφελούνται από τοπικές τιμές. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν πάνε στην Κίνα ή στην Αμερική θα πληρώνουν υψηλή τιμή. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα για το εμπορικό μας ισοζύγιο. Όσον αφορά το διπλό IMSI, τη διπλή διεθνή ταυτότητα κινητού συνδρομητή, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο. Εδώ είμαστε όλοι οι εμπειρογνώμονες για να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τον οικονομικό χώρο για τους παρόχους περιαγωγής, αν έχουμε μια νέα επιχείρηση ως ε, εταιρεία περιαγωγής, πρέπει να αντλήσουμε κεφάλαια, γιατί χρειαζόμαστε τεχνική υποδομή ένα call center και ένα back office. Όλα αυτά είναι δαπανηρά και όταν θα τα έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά πρέπει να προσελκύσουμε και πελάτες με διαφήμιση, θα πρέπει να βρούμε πολιτές, θα τους πληρώνουμε, όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται χρήματα. Ένας πάροχος περιαγωγή που θέλει να ανταγωνιστεί έναν άλλο πάροχο η Vodafone θέλει να ανταγωνιστεί στη Γαλλία παραδείγματος χάρη θα πρέπει η τιμή να είναι 20% πιο κάτω από την τιμή του παρόχου. Αν είσαι μια μικρή εταιρεία όπως η Transatel θα πρέπει να είναι 30% πιο κάτω η τιμή σου. Αυτές οι εκπτώσεις τιμών βασίζονται σε 10 χρόνια πείρας. Μην νομίζετε ότι τώρα κατά τα αναφέρω αυτά τα νούμερα. 10 χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά και ξέρω ότι αν δεν είμαι 30% πιο κάτω από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας δεν πρόκειται να πουλήσω αυτές οι νέες, ε, αυτοί οι νέοι πελάτες που θα βρεθούν σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και πρέπει να καλύψουμε το κόστος κτήσης σε λιγότερο από 12 μήνες για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη επιχείρηση. Σας είπα ποια είναι τα αριθμητικά δεδομένα για την Transatel, χωρίς να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες. Αν δείτε τι διαφορετικές λύσει για το reselling και το dual IMSI, υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Θα δείτε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, ιδίως εάν μειώνεται το ανώτατο όριο για την τιμή λιανικής. Θα πρέπει η Ευρώπη είτε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να περιμένει λίγα χρόνια για να δει ποιε είναι οι επιπτώσει ή να μειώσει το, κόστος, το ανώτατο κόστο τη περιαγωγή. Οπότε δεν θα υπάρχει ανταγωνισμό και θα κλείσουμε σε ένα-δύο χρόνια τη δουλειά μα, την επιχείρησή μα όσον αφορά την περιαγωγή. Η Transatel προσφέρει λύσεις και είναι λύσεις που δουλεύουν στην αγορά. Το έχουμε αποδείξει ότι δουλεύουν. Δεν είναι κάτι το οποίο αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Η δική μας λύση υπάρχει και λειτουργεί. Ούτως ή άλλως ένας εικονικός πάροχος πρέπει να μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες περιαγωγής, γιατί και οι εθνικοί εικονικοί πάροχοι μπορούν να αποτελέσουν ένα παίκτη στο παιχνίδι και αυτό θα έχει επίπτωση στην αγορά. Δεν το έχουμε λάβει υπόψη μέχρι τώρα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επίσης πρέπει να προσέξουμε με τις ρυθμίσεις που θα βάλουμε να μην δώσουμε την ευκαιρία σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες να δίνει καλές τιμές σε πολίτες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή δεν θέλουμε να φεύγουν τα χρήματα από την Ευρώπη και να υποφελούνται οι πολίτες σε άλλες υπήρους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και περνάμε κατευθείαν στον επόμενο ομιλητή, Τόνι Σότελ. Είστε έτοιμος, έχετε και τον υπολογιστή έτοιμο, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπλερ και κύριε Περέλα. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή να απευθύνομαι σε εσά και θέλω να σα ευχαριστήσω και για ω καταναλωτή για τη δουλειά που κάνετε για τι προηγούμενε πρωτοβουλίε για την περιαγωγή. Είμαι και ε, δικαιούχο ε, αυτού του έργου. Ωφελήθηκα όπω και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ο αντιπρόεδρο ε, Κρού μα εξυπηρέτησε όλου θέτοντα φιλόδοξου στόχου το προς ε, το να κινηθούμε μέχρι το 2015 στην εξάλληψη των τελών περιαγωγής, αν όχι μας ε, ανάγκασε όλους ε, να επανεξετάσουμε την προσέγγιση και θέλω να αναφέρω τρία σημεία στο χρόνο που έχω καταρχήν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα διαφορετικό πρόβλημα σε επίπεδο χονδρικής πώληση, όπου βλέπουμε πολλαπλά δίκτυα για, για περιφθοριακή κυκλοφορία. Βλέπουμε να εξελίσσονται ε, πολύ χαμηλά πολύ χαμηλέ τιμέ. Σε αυτή την περίπτωση τη βλέπουμε στο εθνικό επίπεδο, γιατί δεν το βλέπουμε και στη διεθνή περιαγωγή. Πιστεύω ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι ένα θέμα εξισορρόπηση ε, μεταξύ τη ε, κίνηση. Ε, εδώ Βρίσκομαι σήμερα γιατί το 2010 ανέφερα αυτές τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία ως το κύριο πρόβλημα. Μπορώ να αναφέρω τη σελίδα 14 του γράφω εργασία τη Κομισιόν, στο οποίο αναφέρθηκε, το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Οι διαπραγματεύσει κυρίω εξελίσσονται γύρω από το να συμφωνήσουμε μια ισορροπημένη κυκλοφορία και στη συνέχεια να έχουμε ένα περιθωρί, μια περιθωριακή τιμή ε, στην υπόλοιπη κυκλοφορία. Και ενώ η ίδια πραγμάτευση ε, για τη μη κυκλοφορία μπορεί σε ορισμένε ε, περιπτώσει να φτάνει να είναι 40% λιγότερη σε σχέση με το ρυθμισμένο ενότατο όριο. Αυτό ε, δεν φαίνεται στατιστικέ, καθώ το σχετικά, σχετικά μικρό ποσό των μη ισορροπημένων λεπτών μπερδεύεται με τον υψηλό όγκο τη κυκλοφορία που έχει εξισορροπηθεί και η Μπέρεκ είπε ότι μόνο αυτή η πολυπόμενη κυκλοφορία υπόκειται ε, σε ισχυρό ανταγωνισμό. Η συνέπεια είναι ότι οι μικροί παροχοί που έχουν μεγάλο κίνητρο να κερδίσουν ε, την ε, κυκλοφορία σε χοντρική και μπορούν να προσφέρουν χαμηλές τιμές αποκλείονται από την αγορά. Εσείς αναφερθήκατε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κύριε Νίμπλερ στον τομέα των μεταφορών. Θέλω να σας υπενθυμίσω είναι μετερνη... τη γερμανική υπόθεση Εγμετ Creed ε, και Εκεί είχαν ε, απαγορευτεί ε, τα ζεύγη ε, διαδρομών μεταξύ των αερομεταφορέων και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και στην αγορά της περιαγωγής. Ε, εγώ πρότεινα λοιπόν την εξισορρόπηση αυτής της κυκλοφορίας αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν ας το βάλουμε κατά μέρο πολύ συχνά. Οι αγορές της δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα ανταγωνιστικά ανταγωνιστικά αποτελέσματα, όπως τα LUU ή τα MTRs. Έτσι λοιπόν όταν δεν είναι ανταγωνιστικά η ρύθμιση προσπαθεί να θέσει τιμές που ε, να προσεγγίζουν το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα και προστατεύουν στους κατανοητέ, υποθέτω ότι υπάρχει επαρκή ανταγωνισμό, έτσι ώστε ε, να έχουμε και χαμηλές τιμές και Πιστεύω ότι η Μπέρεκ έχει κάνει ε, ηρωικό έργο στο να εκτιμήσει το κόστος ε, στην περιαγωγή αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι τα δεδομένα ήταν πολύ περιορισμένα. Επίση είπαν ότι τα αποτελέσματά του είναι πολύ συντηρητικά. Πιστεύω ότι το κόστο που έχει το πιστεί υπερδηλώνει το κόστος της χονδρικής ε, και ήδη έχουμε έναν αριθμό παρόχων που να προσφέρουν ε, τιμές ε, χονδρικής μεταξύ 1 και 5 λεπτών 1 μεγαμπάιτ. Έτσι λοιπόν σήμερα στην Πολωνία την προσφέρει ένα 10 ευρώ ανά γιγαμπάιτ ανοιχτό στην αγορά σε τακτική βάση. Ε, τρέχουν όλοι για να εκμεταλλευτούν ε, αυτή τη φανταστική τιμή ή όχι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ισορροπίας, αλλά υπάρχουν πολλές συμφωνίες με διάφορους παρόχους ε, στα 5 λεπτά ένα μεγαπάιτ και βλέπω ότι ορισμένοι από τους παρόχους βρίσκονται εδώ σήμερα. Τώρα, για να να μιλήσουμε για ποσοστά, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι υπάρχει στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, για τι συγχετικέ ε, συνομιλίε ε, και τα SMS, νομίζω ότι η κυρία Νίμπλερ έρχεται πιο κοντά σε κάτι που ε, προσεγγίζει το κόστο. Ε, Όμω, ακόμη και αυτό είναι χαμηλότερο μέσα στο βεληνικέ ε, κόστου τη Μπέρεκ αν ε, οι τιμές ε, της ε, χονδρικής προσεγγίζουν το κόστο, τότε θα πρέπει να είναι προσφέρουν να κάνουμε μια πανευρωπαϊκή προσφορά σε γενικό επίπεδο. Αυτό ήταν ο αρχικό κόστο που θέτηκε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό μέσα σε ορισμένα όρια. Αν δούμε την αγορά στι ΗΠΑ, οι παναμερικές προσφορές είναι περιορισμένε. Κανένα παρέχο στι ΗΠΑ δεν έχει παναμερικανικό δίκτυο. Όλοι χρησιμοποιούν υπηρεσίε περιαγωγή σε μικρότερο σε μεγαλύτερο βαθμό και σίγουρα οι υπόλοιποι παροχοί πέρα από τους τέσσερις σε μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τέσσερι κυρίες παροχής της ΕΠΑ έχουν συμβατικούς περιορισμούς ε, αν πριν το σχάρι συνεχώς ε, βγαίνει από το δίκτυό σου τότε κάποια στιγμή θα, θα υπάρχουν θα υπάρχουν περικοπές. Εμείς όμως ε, πρέπει να δούμε το σύνολο της ε, τιμής χονδρικής. Πρέπει να τεθεί σε κατάλληλο επίπεδο. Έχουμε μόνο μία λύση να προτείνουμε που είναι τα τα όρια τιμών. Σε χονδρικό επίπεδο όμως έχουμε δύο ανταγωνιστικές, τιμές, ε, δύο ανταγωνιστικές λύσεις να προτείνουμε σε επίπεδο λιανικής. Τα διαφορετικά μέτρα που προτείνονται προτείνονται μόνο για να περάσουμε ε, από τα νότα χονδρική στο λιανικό επίπεδο. Όμως ε, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των πολύ χαμηλών ε, τιμών λιανικής Όπω είπε και ο κύριο Απτιτρεζατέλ, έναντι του να θέσουμε πάρα πολύ υψηλέ τιμέ ελληνική και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως στόχος, της αγορά, συγγνώμη, ως στόχος τιμών στην αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να αφαιθεί επαρκής χώρος ε, μεταξύ των δύο τιμών ε, ε, στη Λιανική και στη Χονδρική για να επιτρέψουμε την είσοδο των νέων παρόχων και έτσι θα δούμε μια ανταγωνιστική διαδικασία μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Τώρα, τα ανώτατα τιμών είναι κατάλληλα για να επιτρέψουν ε, να λειτουργήσουν τα διευθυντικά μέτρα. Έτσι όπως προτάθηκε ο κανονισμός κομισιών θα μπορούσε να αποσυρθεί αν δεν εξελιχθεί ο ανταγωνισμός είτε μεταξύ των υφιστάμενων ε, παρόχων ε, είτε με καινούριων είναι δυνατό να επανεισάγουμε χαμηλότερων τιμών μετά το 2016 και υποπτεύουμε ότι κανένας δεν θα ανέμενε αυτό τον οίκο να είναι και πάρα πολύ μαλτακός σε αυτή την προσέγγιση. Δεδομένης της περιορισμένης φιλοδοξίας των διευθυντικών μέτρων, Δηλαδή να περάσουμε από το κόστος της, της χοντρικής στη το κόστος και η ταχύτητα της εφαρμογής ε, είναι σημαντικές πτυχές ε, και νομίζω η λύση ενός ε, και μόνο λύση είναι η καλύτερη. Ε, ενός και μιας και μόνης διεθνής ταυτότητας ε, κινητού συνδρομητή δηλαδή. Ε, νομίζω ότι θα, πρέ... θα μπορούσαμε να πετύχουμε, θα, πρέπει να θέσουμε το στόχο μιας πανευρωπαϊκής προσφοράς και να θέσουμε τη μέση πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Μόνικα Σταρναρόβα. Ελπίζω να πρόφερα σωστά το δύσκολο όνομά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις κυρίες Ένιμπλερ και Κόρχολα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στην σημερινή ακρόαση για να σας πω ποιες είναι οι δικές μας απόψεις για την πρόταση σε ό,τι αφορά ε, την περιαγωγή. Μια πρόταση πάρα πολύ σημαντική για τις, ε, για της περιαγωγής είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που τυχόν θέλετε να θέσετε και εσείς και θα επικεντρωθώ στην ομιλία μου στη σκοπιά του καταναλωτή. Αλλά καταρχάς σας δώσω μια γενικότερη εικόνα. Μεγάλη κινητικότητα σήμερα, έχουμε μεταφορά φωνής και δεδομένων ε, που προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία μέσα στι υπηρεσίε. Οι τιμέ της περιαγωγή είναι υψηλέ και παραμένουν εμπόδιο. Αν δούμε την ίδια την έννοια του roaming, της περιαγωγή δείχνει ξεκάθαρα νομίζω ότι εδώ η αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει τεχνική αιτιολόγηση για να παραμένει έτσι η κατάσταση. Αν δει κανεί τι αγορέ τώρα, 4,5 χρόνια μετά την ε, θέση σε ισχύ ε, του κανονισμού περιαγωγή 1, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, εξακολουθούν να βλέπουν ότι χρεώνονται πολύ ψηλέ τιμές για τις υπηρεσίες περιαγωγής και οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται και δεν χρησιμοποιούν τα κινητά τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μάλιστα προτιμούν και να τα απενεργοποιήσουν εντελώς για να μην τους έρθουν υψηλοί λογαριασμοί. Αυτό το έδειξε και το Ευρωβάρομετρο από το 2010 που ήταν αφιερωμένο στην περιαγωγή. Τώρα, πώς θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω θα πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια για τις διασυνορικές δραστηριότητες, να, είναι πιο, ε, να νιώθουν πιο ασφαλείς οι καταναλωτές, να χρησιμοποιήσουν εξωτερικό τα κινητά τους. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για ένα νέο κανονισμό για την περιαγωγή. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να καταργήσουμε κάποιες από τις χρεώσεις ε, της περιαγωγής και να είμαστε δηλαδή πιο προβλεπτικοί. Θεωρούμε αυτόν τον νέο κανονισμό ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά βήμα στην κατεύθυνση ε, μιας Ευρώπης από το roaming. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποδεσμοποίηση, δεν ε, θα συζητήσω για τις λύσεις για να σας πω ποια είναι η καλύτερη. Εν γέννη πιστεύουμε ότι η αποδεσμοποίηση με την χονδρική πρόσβαση στο roaming και η υποχρέωση για μη διακρίση θα μπορούσε να βελτιώσει σε κάποιο βαθμό τον ανταγωνισμό, αλλά και να ε, φέρει νέες προσφορές για υπηρεσίες περιαγωγής που βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, να υπάρχει τέτοια ανάγκη, ιδίω ε, στην κυκλοφορία των δεδομένων που αυξάνεται. Η πρόταση η ε, θα πρέπει να βασίζεται σε μια ουδέτερη από τεχνολογική πλευρά προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτά που προτείνει και η κυρία Νίπλε στην εκθεσή τη. Θα πρέπει δηλαδή μόνο οι βασικέ αρχέ να υπάρχουν. Κάθε τεχνική ε, λύση, δηλαδή τι αρχέ πρέπει να πληρεί. Οι βασικές αρχές κατ' είναι η τεχνική λύση να είναι αποδοτική, να είναι φιλική προς το χρήστη και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενημέρωση των καταναλωτών, πώς θα νιώθουν πιο ε, μεγάλη εμπιστοσύνη και θα χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες περιαγωγής καταναλωτές. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η αποδεσμοποίηση θα φέρει νέα στοιχεία για τους καταναλωτές, θα απαιτήσει και την αλλαγή των συνηθιών των καταναλωτών σε κάποιο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση προς τους καταναλωτές για το ότι μπορούν να επιλέξουν ένα αλλακτικό πάροχο αλλά και να είναι σαφείς εύληπτες και διαφανείς πληροφορίες που θα λαμβάνουν καταναλωτές ό,τι αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών για να μην, υπάρχουν, ε, για να μην υπάρχει παραπλάνηση των καταναλωτών. Είναι ξεκάθαρη η όροι, σαφέστατη. Σε ό,τι αφορά επίση τη διαφήμιση θα πρέπει να τηρείται πλήρωση η νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, ιδίω ό,τι αφορά την οδηγία της αθέμητη εμπορική πρακτικές. Τώρα, ρύθμιση των τιμών. Όπως είπα, η αποδεσμοποίηση εγγυάται την πρόσβαση ε, στην περιαγωγή και μπορεί αυτό να είναι θετικό για τον ανταγωνισμό και να φέρει νέες ε, εναλλακτικέ λύσει. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εξακολουθεί να παραμένει απαραίτητη η ρύθμιση των τιμών. Υπάρχει μια ειδική πρόταση για τη ρύθμιση των τιμών. Σε ό,τι αφορά τις ε, φωνητικές υπηρεσίες ή και εν γέννη για τις υπηρεσίες ε, roaming, θεωρούμε ότι θα πρέπει να, η τιμή για τον καταναλωτή να είναι προσανατολισμένη περισσότερο προς το κόστος. Σε ό,τι αφορά ε, τη φωνή, να αναφέρω τα εξή στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε οι χρεώσεις να ευθυγραμμιστούν με τις εθνικές τιμές μέχρι το 2015, Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε με τα 15 cent σωστά το τιμή. Από το 2012 ήδη και μετά να μειωθεί στα 13 και να φτάσει στα 10. Αν δούμε τώρα το scoreboard για το 2011, θα δούμε ότι η μέση τιμή το λεπτό για, τις, για την κινητή επικοινωνία ε, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 ήταν 13 cents, το 2009 ήταν 10 cents. Για το 2011 δεν έχουμε αποτελέσματα, αλλά μπορούμε να περιμένουμε χαμηλότερη τιμή. Άρα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τις τιμές ε, για τη φωνή. Τόσο ότι αυτά τα SMS, υπηρεσίες περιεγωγής, πάλι προσανατολισμένες προς το κόστος. Αν δει κανείς την τιμή για την παροχή της υπηρεσίας, ένα με δύο cents είναι περιοχή των τιμών. Και αν δούμε τα ανώτατα όρια που είναι γύρω στα 10 cents. Γιατί, γιατί δεν χρησιμοποιείται συχνά υπηρεσία. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπάρχει τόσο τεράστιο περιθώριο. Προτείνουμε λοιπόν 7 cents. Ως ε, αφετηρία. Το 2012 δηλαδή. Τώρα στα δεδομένα. επικροτούμε την πρόταση της Κομισιόν να έχει ανώτερες τιμές ε, λιανικής ε, για αυτές τις υπηρεσίες, μεταφράζω στην περιαγωγή, αλλά θεωρούμε πολύ υψηλή την τιμή ανά μεγαμπάιτ. Σε κάποιες χώρες βρίσκουμε και τιμές της τάξης του 5, των 5 cents. Γιατί 19 λοιπόν εδώ. Καλά, καλό είναι να έχουμε ένα περιθώριο για την αποδεσμοποίηση, αλλά το περιθώριο 100% νομίζουμε ότι είναι κατάλληλο. Τελευταίο σημείο. Διαφάνεια και αναθεώρηση. Με τις σημερινές διατάξεις ε, προστατεύονται οι καταναλωτές. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όταν, όταν ταξιδεύουν εντό ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να είναι πλήρως προστατευμένοι και καλυπτόμενοι ε, και να μην έχουν τέτοια προβλήματα, να πάθουν σοκ βλέποντας έναν υψηλό λογαριασμό, θα πρέπει να καλύπτονται και τα SMS. Και αυτό θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση για τις υπηρεσίε Ρώμη. Και για αυτού που προπληρώνουν και για που πληρώνουν εκ των υστέρων. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τώρα, Σε ό,τι αφορά τώρα την υλοποίηση της αποδεσμοποίησης, αν αποφασιστεί να εφαρμοστεί αυτό, ίσως είναι πρόημο να γίνει Θεός το 2015. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων αυτών των διορθωτικών μέτρων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εκτιμήσει πάρα πολύ προσεκτικά τη λειτουργία της αγοράς. Λειτουργεί αποδοτικά, να το δει το 2016 ίσως αυτό και αν όχι να προτείνει κάποιες περαιτέρω λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Χάρμπορ και εσείς. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους. Και τώρα θα έχουν οι συνάδελφοι την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις. Παρακαλώ να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικοί, να είμαστε σύντομοι και ακριβεί. Ο κύριος Παύλου Γουμπι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για την αρχή του must carry θέλω να ρωτήσω. Κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών ε, τι συμβάσεις μπορεί να έχει και πώς μπορούμε να έχουμε κάποια σχετική ρύθμιση των τιμών. Άλλη ερώτηση. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Κριστίαν Έγκστρομ. Ε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Μούρικ τη τηλεφώνικα. Είπατε ότι συμφωνείτε με τις ανώτατες τιμές της Επιτροπής. Ε, ε, οι τιμές χονδρικής είναι 300, 200 και 100 ε, που και μειώνονται συνεχώς ως ανώτατα όρια χονδρικής. Εγώ θα πρότεινα 10 ευρώ ανά μεγαμπάιτ. Και το έχω συζητήσει και με άλλους εκπροσώπους της τηλεφώνικα φάνηκε ότι δεν είναι, από τη λένε δεν είναι λογική η τιμή. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν είναι λογική μια, ένα ανώτατο όριο τιμών 10 ευρώ, γιατί δεν είναι λογικό. Η κυρία Νίμπλερ είπε ότι ήταν 8,80 η τιμή ηλιανική στη Γερμανία. Η τηλεφώνικα μπορεί να προσφέρει και κάτι καλύτερο στους Ισπανούς καταναλωτές. Εσείς προσφέρετε 2 GB το μήνα για 12,5 ευρώ. Δηλαδή 6,25 ευρώ ένα γιγαμπάιτ. Αυτή είναι η τιμή νικής προς τους Ισπανούς καταναλωτές. Αν μπορείτε να το προσφέρετε λοιπόν στους Ισπανούς καταναλωτές με 6,25, γιατί θεωρείτε τα 10 ευρώ ως παράλογο ανώτατο όριο. Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις με πολλές διαφορετικές απόψεις ανάλογα με την προέλευσή τους κάθε φορά. Σχετικά με την έννοια του ανωτάτου ορίου που θα έπρεπε να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στα εγχώρια όρια. Υπάρχει ενδεχομένω ένας κίνδυνος τα τέλη περιαγωγή να βασίζονται στα εγχώρια τέλη και ε, τα καρτέλ να υποφεληθούν. Όταν πρωτοβάλαμε ανώτατο όριο, θυμάστε ότι μας πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα το χειριστούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεκαστήγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι Έχουμε δραματική μείωση των τιμών ε, σε επίπεδο ε, γιατί μιλάμε εκ μέρους του καταναλωτή στην αγορά περιαγωγής. Όμω, ε, πολλέ φορέ όταν σκεφτούμε έναν χώριο παροχό φαίνεται να πιστεύουν όλοι ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν αν πάνε τα πράγματα προ το να έχουμε κάτι παρομοίο με τις εγχώριε τιμέ, αυτό θα ήταν καλό. Θέλω να ρωτήσω τον πρώτο μιλητή που εκπροσωπούσε την τηλεφώνικα, τον κύριο Μούρεκ. Μήπω μπορείτε να μα αναφέρετε κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε ε, σε σχέση με αυτή την εναλλακτική του Near Domestic Pricing, ε, δηλαδή επί της αρχής, ξέρετε, ακούγεται ελκυστικό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω λεπτομέρειες και περαιτέρω εκπόνηση αυτού του θέματος. Ο κ. Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές, τους προσκεκλημένους σήμερα το απόγευμα. Καταρχήν να πω ότι ορισμένα από τα σχόλια που άκουσα ορισμένες από τις προτάσεις ε, στην πρόταση της Κομισιόν ακούγονται αρκετά πολύπλοκα για μένα. Και ε, πραγματικά ε, φαίνεται να υπερισχύεται το επιχείρημα εξφορτής με την όλη διαδικασία. Αυτό ήταν το πρώτο που θέλω να πω. Και να πω ότι με ελκύει η πρόταση να έχουμε εξαίρεση για τους παρόχους που χρεώνουν ε, τιμές κοντινές ε, στις εγχώριες χρεώσεις. Ε, γιατί τελικά στο δύο καταλήγουμε, το να ξεφορτωθούμε. Επίσης, το ότι δεν μου αρέσει καθόλου είναι παραδείγματο χάρη ε, το ότι εμείς χρεωνόμαστε γιατί λαμβάνουμε αυτές ε, τις ε, κλήσεις και κάποιοι είχαν προτείνει να μην υπάρχει καμία χρέωση για τις κλήσεις που λαμβάνουμε. Θα επανέλθουμε όμως να σας πω ότι πραγματικά με ανησυχεί κάποιοι που είπατε ότι σας αρέσει η πρόταση Κομισιόν και χρησιμοποιείτε τον κλάδο. Όμως ε, θα ήθελα να σας πω, ακούσαμε ορισμένε προτάσεις για το πώς εμείς ως νομοθέτες μπορούμε να αντικοποιήσουμε τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό χωρίς ε, να μπούμε στη μικροδιαχείριση των ανώτατων ορίων τιμών και των κατοφυλιών. Γιατί εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιες λύσεις από τον κλάδο. αν ε, μπορείτε να ασκήσετε τις δεξιότητές σας, είτε αυτές είναι επιχειρηματικές είτε τεχνολογικές, προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ έχω δύο-τρεις ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες όσον αφορά τα διαρθρωτικά μέσα. Ακούγοντα και αυτά που είπαν οι ομιλητέ και ο Τζέλ Σίτσεστερ, μερικέ φορέ ε, μπερδεύομαι περισσότερα. Σχετικά με το «Must Carry». Το είπε και ο εκπρόσωπο τη Τρανζατέλ. Είπατε και εσεί ότι δυσκολευτήκατε να συνάψετε συμφωνίε περιαγωγή. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίε στη σύνεψη συμφωνιών ε, περιαγωγή. Πολύ συχνά υπάρχει το μάσκαρι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στην αγορά όπου θέλει κανείς να έχει πρόσβαση. Ο συνάδελφος, ε, ο κύριος Μουρίκα από την Τελεφώνικα, ε, είπε ότι καταρχήν συμφωνεί με ε, τα διαστατικά μέσα και πρέπει να δούμε τα περιθώρια τιμής. Ο κύριος Φόρες διαφωνεί με τα διαρθρωτικά μέτρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι οι ομιλητές ε, έχουν διαφορετικές απόψεις. Καταλαβαίνετε πόσο δυσκολευόμαστε και εμείς ως νομοθέτες να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα τεχνικά μέσα είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ε, ενιαίο ύμση, το διτό ύμση, είναι τόσο πολλά τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε που καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι ο τομέα. Μετά από τον κύκλο των ομιλητών που ακούσαμε, μου κάνει όλο και μεγαλύτερη εντύπωση πόσο πολλές διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Είναι δύσκολο λοιπόν το έργο μας σε σχέση με αυτό το θέμα και κλείνοντας επανέρχομαι σε αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος Τσίσεστερ. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ε, δεύτερο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Δεν άκουσα να λέγεται κάτι για τις εγχώριες τιμές. Πώς μπορούμε για τις εγχώριες τιμές ε, να έχουμε τόσο καλές προσφορές και με το που περνάμε τα σύνορα να έχουμε πλάσεις και 30 φορές παραπάνω τιμές. Δεν νομίζω ότι είναι λογική αυτή η τακτική. Γιατί να είναι έτσι. Μπορούμε ε, να καταλήξουμε σε κάποια λογική τιμή, σε κάποια εξισορρόπηση, αυτό το balancing που αναφέρατε, για να είναι η κατάσταση αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Κορόλα. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι πολλές φορές ανέφεραν ε, αυτές τι φανταστικές εγχώριε προσφορές ε, και ρώτησε μου στους παρόχους είναι Είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι εγχώριες ε, προσφορές αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος ή μπορεί να είναι τόσο δυνές απλώ επειδή οι πάροχοι εταιρείε καλύπτουν το κόστος μέσω των κερδών ή των περιθωρίων κέρδους που λαμβάνουν από την περιαγωγή. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Ίσως θα μπορούσατε να απαντήσετε όμως σε αυτό. So, wir jetzt mal eine Ας κάνουμε και ένα γύρο απαντήσεων, να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν στις μέχρι τώρα ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά, όπως σας βλέπω εγώ, και με τη σειρά θα απαντήσουν όλοι οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Ρομπέρτ Μούρικα από την Πεντελεφώνικα. Μου απευθύναν κάποιε ερωτήσει σε μένα προσωπικά. Να απαντήσω σε αυτά καταρχήν λοιπόν. Υπήρχε μια ερώτηση γιατί το όριο, το ανώτατο όριο τιμής ε, για τα δεδομένα ήταν τόσο ψηλό. Ειλικρινά. Η περιαγωγή δεδομένων είναι αρκετά ακριβή και νομίζω ότι όλοι οι πάροχοι το έχουν αναγνωρίσει αυτό και βλέπετε ότι υπάρχει αλλαγή στην αγορά αυτή τη στιγμή. Μειώνονται σχετικά γρήγορα οι τιμές ε, για το roaming, περίπου 50%. Ετησίω έτσι λοιπόν ο ανταγωνισμός σε αυτή την αγορά αρχίζει να λειτουργεί. Και γιατί αρχίζει να λειτουργεί, γιατί Πολλοί πελάτες τώρα έχουν ε, smartphones και θέλουμε ε, να ε, πείσουμε στους να αρχίσουν να αλλάξουν αυτά τα smartphones και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους. Και αν μειώσουμε την τιμή, δεν βλέπουμε ε, αυξημένη χρήση για τη φωνή, ενώ με τα δεδομένα για τις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ ισχύει το αντίθετο με τα δεδομένα, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη χρήση αν μειωθεί η τιμή. Γι' αυτό αντιδρά λοιπόν η αγορά και κάνει ακριβώς αυτό που απαιτείται. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει εν μία νυχτή. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται σταδιακά. Και όπως είπα, νομίζω ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα τιμών τα οποία όλοι ελπίζετε σύν το χρόνο, αλλά αν δώσετε μία ευκαιρία στην αγορά θα προχωρήσει βήμα το βήμα και θα έχουμε φτάσει εκεί μέχρι το 2015. Τώρα, ποιο είναι το πραγματικό κόστος των δεδομένων, δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν ε, διάφορα προϊόντα δεδομένων, ε, από μηχανή σε μηχανή, ε, το χάρη και αυτό είναι πιο ακριβό από μακρές ροές δεδομένων. Εξαρτάται λοιπόν από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί κανείς και το, από το είδος των υπηρεσιών αλλά νομίζω ότι οι τιμές οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχω μια ερώτηση από την κυρία Πιλάρδο Καστίγιο για αυτή τη λύση του Near Domestic Pricing. Εδώ, τι έχουμε κατά νου. Δεν το έχουμε προσδιορίσει ακριβώς αυτό. Εμείς έχουμε κατά νου κάτι παρόμοιο που ανέφερε ο συνάδελφος από την Μπουίκ. Δεν ε, έχουμε κάποιους τύπους που θα εφεύρουν οι ε, πάροχοι για να... Μάλλον υπάρχουν κάποιες τέτοιες φόρμουλες που θα μπορούσαν να εφεύρουν οι για να δώσουν κάποιες τιμές ε, που να είναι πιο κοντά στην χώρα παραγωγή. Παραδείγματο χάρη για ένα ευρώ την ημέρα θα μπορούσε κάποιο ε, να έχει όσο περιεχογή θέλει τέτοιου είδου λύσει. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις ε, φόρμουλες ε, λιανικής ε, που μπορούν να εμπνευστούν οι πάροχοι, αλλά ίσως θα πρέπει η Μπέρεκ να μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το τι σημαίνει αυτό το near domestic και τι εμπίπτει σε αυτές τις παραμέτρους. Και αν ένας πάροχο πράξει αυτό, τότε έχουμε ανταγωνισμό και από ένα εγχώριο πάροχο, δηλαδή ένα ισπανικό, ένας ισπανικός πάροχος παρέχει ε, τέτοιες τιμές και έτσι λοιπόν ασκείται πίεση στις άλλες εταιρείες τις ισπανικές να παρουσιάσουν καλύτερες τιμές βάσει της διευθυντικής λύσης ή να κάνουν κάτι παρόμοιο. Έτσι λοιπόν, ε, με αυτόν τον τρόπο εισάγεται ανταγωνισμό στην αγορά. Όμω οι ίδιοι οι πάροχοι πρέπει να αποφασίσουν αν επιθυμούν διαφορετική λύση ή κάτι που μπορούσαμε να το αποκαλούσαμε near domestic price. Γιατί λέω near domestic, γιατί υπάρχει κόστο. και πάντοτε θα υπάρχει κάποιο κόστο στην περιαγωγή. Ο κύριο Τσίτσεστερ ε, αναφέρθηκε στι κλήσει που λαμβάνουμε. Νομίζω ότι ε, στην περίπτωση αυτή υπάρχει κόστος και αν ε, υλοποιήσετε κάποιες από τις φόρμουλες που ανέφερα, θα μπορούσατε απλώς ε, να ανακτήσετε το και να καλύψετε το κόστος αυτό. Η κυρία Νίμπλερ ε, ρώτησε γιατί χρειάζομαι περισσότερο για την περιαγωγή. Κατά τη δική μου εμπειρία, η απάντηση είναι οικονομικού χαρακτήρα και έχει να κάνει με την ελαστικότητα των τιμών. Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά αν ε, ρωτήσετε ένα πελάτη τι θέλεις, πολύ φτηνά, πολύ φτηνές τιμές ε, στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θα πληρώσεις ε, περιαγωγή, θα πληρώσεις πιο ψηλές τιμές στο εγχώριο επίπεδο, αλλά δεν θα πληρώσεις περιαγωγή, οι περισσότεροι θα επιλέξουν τα πολύ χαμηλές τιμές στο εσωτερικό επίπεδο. Εκεί βρίσκεται ο ανταγωνισμός και ως πάροχος επιλέγεις ε, να θέσεις κάποιες λογικές τιμές θέτοντας επιπλέον κόστος στην περιεγωγή. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από την BUIG. Ε, θέλω να συμπληρώσω ότι είπε ο συνάδελφο για ποιο λόγο είναι τόσο υψηλέ ε, οι τιμέ περιαγωγή. Νομίζω ότι ε, προέρχεται από τον κόσμο των κινητών, από το κόστος ε, ενό λεπτού ε, κλήσης ήταν πολύ ψηλός και το business model της περιαγωγής βασίστηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις και κατόπιν στο SMS και στο Megabyte. Με τις νέες τεχνολογίες, το ριζόνι που είναι διαθέσιμο για τους πελάτες είναι ευρύτερη, όλο ένα και μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να πείσουμε ε, την Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχουμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που να λαμβάνει υπόψη τι πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. Ε, Παραδείγματο χάρη ένα καταναλωτής στη Γαλλία ε, έχει ευρεία κάλυψη και πληρώνει περισσότερο και παραδείγματο χάρη μπορεί να πληρώνει λιγότερο για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Ενώ θα πρέπει να πληρώσει για το γεγονό ότι δεν έχει παραδείγματο χάρη πληρώσει για Ευρωπαϊκό Δίκτυο, δεν έχουν γίνει πρόσθετες απαιτήσει και όχι τόσο για τα πρόσθετα λεπτά. Γιατί ε, δεν θα βαρύνει το δίκτυο αυτό και στις χώρες περιεγωγής ε, θα υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ε, ε, υψηλών χρηστών και των μικρότερων χρηστών. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι αυτό το πρόσθετο τέλος για τη γεωγραφική επέκταση Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ο Γάλλο καταναλωτή ε, δεν ε, έχει πληρώσει για ένα γερμανικό ή για ένα λοδίκτυο και έχει ένα προ το τέλο να πληρώσει. Παραδείγματο χάρη, ένα ευρώ την ημέρα και αν αγοράσει ένα ολόκληρο μήνα, ε, τότε θα πληρώνει λιγότερο από 30 ευρώ, γιατί αυτό θα είναι συνδεδεμένο. Και θα υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων παρόχων και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καλύτερο τρόπο να εφαρμόσουμε του στόχου του ψηφιακού θεματολογίου. Δηλαδή να μην ε, έχουμε την ίδια τιμή σε χώριο επίπεδο και τιμή περιαγωγής ε, και τελικά δεν ε, θα υπάρχουν δεν θα υπάρχει πλέον επίπεδα τιμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περιεγωγή 1 και στην περιεγωγή 2 είχαμε ρυθμισμένε τιμές και δεν υπήρχε κίνητρο για την πρόθεση του ανταγωνισμού γιατί μετά από το roaming 1 και roaming 2 ε, εγώ μετέβη σε διάφορες ε, χώρες ε, και είπα δώστε μου τοπική πρόσβαση έτσι ώστε να μπορέσω να αναπτύξω την επιχείρησή μου στη χώρα σας και υπήρχαν άνθρωποι ενώπιον μου που θεώρησαν ότι δεν ήταν η κατάλληλη να μειώσουν την πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα το Roaming 3 διαφέρει γιατί ο όρος ανταγωνισμός είναι στο κείμενο για πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να αποφασίσουμε είτε θα βάλουμε ως προτεραιότητα να προωθήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό και πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό για να λάβει χώρα αυτός ο ανταγωνισμός, τουλάχιστον δύο χρόνια θα έλεγα, και κατόπιν δεν ε, μπορείτε να είστε πολύ αυστηροί στο νοτοτορείο της περιαγωγής γιατί θα σκοτώσετε τον ανταγωνισμό και μάλιστα το 2012 ξέρετε από δημοσιονομική σκοπιά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα ή θα πείτε δεν θέλουμε ανταγωνισμό και θέλουμε τοπική τιμή οπουδήποτε και να κάνει στην Ευρώπη, γιατί όχι, αλλά αυτή είναι πολιτική απόφαση. Αλλά δεν ε, προσφύμαστε εδώ ότι θέλουμε ανταγωνισμό, ή το ένα ή το άλλο. Αλλά αν θέλουμε ανταγωνισμό, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο σε εταιρείε όπω τη δική μου. Εάν κάποιο άλλο θέλει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να προσπαθήσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Ευχαριστώ. So, um σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου Τσίτσεστερ και το ερώτημα της κυρίας Νίμπλερ για τον ανταγωνισμό. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Τρανζατέλ ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον ανταγωνισμό να πετύχει. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε χώρο μεταξύ των ε, επιπέδων τιμών λιανικής και των άτομων τιμών χονδρικής. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε τον ανταγωνισμό στο επίπεδο το λιανικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση οποιοδήποτε μέτρου που θα εισήγαγε ανταγωνισμό σε επίπεδο χονδρικής. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή και είναι και ενδιαφέρον με ένα-δύο ποσοστό διαφορετικό βλέπουμε ότι οι εταιρείε ε, που έχουν ένα μεγάλο ε, ποσοστό παρέχουν και σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά αυτό ε, δεν είναι λογικό γιατί καθένας πάροχος θα μπορούσε να παρέχει τις υπηρεσίες και αυτό μειώνει τον, το πεδίο για τον ανταγωνισμό. Ένα μικρό σχόλιο, αν με επιτρέπετε, για αυτό που είπατε, ανταγωνισμός, ανώτατα όρια. Νομίζω ότι με χαμηλότερα όρια πάλι μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό. Ποιο είναι το δίκαιο περιθώριο εδώ, fair margin. Ώρες θα μπορούσαμε να το συζητάμε. Αυτό το 100% ήδη είναι αρκετό, είναι πολύ. Άρα νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός και με αυτό το ποσοστό. Ένα μικρό σχόλιο. Ή εγώ έχω συστήσει το 2000 ε, την εταιρεία μου με την αρχή του Ρώμη και ήταν μια εταιρεία αρμπιτράς και πλήρωσα 1.800 ευρώ για δύο χρόνια. Πριν έβγαζα χρήματα ήμουν και στη Μακένζη σύμβουλος. Δεν είναι όμως εύκολο. Εντάξει να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει περιθώριο. Υπάρχει αλλά Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι τέτοιες δηλώσεις του αέρα. Πρέπει να έχουμε στοιχεία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νίμπλετ από τον ε, Μπέρεκ, από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Αν θέλετε βέβαια να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε τον Μπέρεκ ε, να συμμετάσχει. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για λίγα μόνο σημεία από τα πάρα πολλά που αναφέρθηκαν. Ξεκινώντα από τον ε, Τόλι Σόρτολ για το θέμα ε, του κόστου χονδρική. Ε, είπατε ότι είναι ηρωικέ οι προσπάθειε τη Ένωση Μπέρεκ. Δεν μα έχουν ξαναπεί οι ήρωες και με τιμά πολύ ο χαρακτηρισμό σα. Είπατε ότι είναι συντηρητικέ οι εκτιμήσει του Μπέρεκ. Οι καλύτερε εκτιμήσει που θα μπορούσαμε να κάνουμε με τα στοιχεία που είχαμε, αυτέ ήταν. Ακούγοντας ε, τα σχετικά με την τιμολόγηση λιανικής σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα δεδομένα, ίσως καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι την επόμενη φορά ο Μπέρεκ θα πρέπει να αναθεωρήσει τα στοιχεία του, παίρνοντα μοντέλα κόστους πιο επικαιροποιημένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια μοντέλα, σε μια-δυο χώρες μόνο έχουμε. Νομίζω ότι τα τελικά μας στοιχεία θα είναι ακόμη πιο χαμηλά από αυτά που είχαμε την προηγούμενη φορά. Εντύπωσή μου είναι βέβαια, δεν έχω κάτι να το στηρίξω αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία πάντως που βάλαμε τα βασίσαμε στις καλύτερες εκτιμήσεις που είχαμε διαθέσιμες. Ο Τόνι συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του αν μειωθούν ε, τα στοιχεία κόστου σημαντικά θα αρχίσουν οι εταιρείε να προσφέρουν πανευρωπαϊκές τιμές, τιμές όπου η τιμή περιαγωγή θα είναι λίγο πολύ ίδια όπως και οι υπηρεσίες οι εγχώριες. Θα συμβεί κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω. Αλλά μέχρι να μειωθούν σημαντικά οι τιμές χονδρικής αποκλείεται να γίνει. Άρα είναι προϋπόθεση η μείωση των τιμών χονδρικής για να επιτύχουμε τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου. Και ίσως οι τιμές πρέπει να πέσουν ε, όσο αυτό που προτείνει η κυρία Νίμπλερ ως ανώτατα όρια ή και ακόμη χαμηλότερα μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό στις τιμές λιανικής, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα διαρθρωτικά μέσα είναι ένας τρόπος βελτίωσης του ανταγωνισμού, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Εάν έχουμε τέτοιες πανευρωπαϊκές τιμές, που θα προσφέρονται από κάποιους που θέλουν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και βλέπουν μια ευκαιρία στο να προσφέρουν πανευρωπαϊκές τιμές, αυτό θα ήταν ένας τρόπος να μπει ο ανταγωνισμός στην αγορά αυτή, δημιουργώντας ανταγωνισμό στην αγορά περιαγωγής, κάτι που βλέπουμε πολλές φορές σε μεμονωμένες χώρες. Η κυρία Νίμπλερ έκανε μια ερώτηση για τις τιμές περιαγωγής. Γιατί είναι τόσο υψηλές ε, οι τιμές ε, περιαγωγής. Ο κύριος Μούρικ έδωσε μια απάντηση οικονομολόγου. Εγώ θα σας δώσω μια πολύ απλή απάντηση. Είναι πολύ ψηλέ οι τιμές περιαγωγής, ε, διότι οι εταιρείε μπορούν να το κάνουν. Δεν υπάρχει πίεση και μπορούν να έχουν πολύ ψηλά τις τιμές τους. Και όσο δεν υπάρχει ανταγωνιστική πίεση, θα συνεχίσουν να έχουν πολύ ψηλέ τιμές. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μειωθούν οι τιμές είναι να ασκηθεί πίεση. Όσον αφορά αυτό το δίλημα που ανέφεραν αρκετοί οι ευρωβουλευτές και κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες, δηλαδή ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των τιμών, είναι ένα θέμα πολιτικής. Ο Μπέρεκ είναι υπέρ του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε μπορούμε να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό, χωρίς να είμαστε δογματικοί ο ανταγωνισμός είναι ένα μέσο προς την επίτευξη του στόχου. Δεν είναι αυτός σκοπός ο ανταγωνισμός. Θέλουμε να έχουμε καλές τιμές και καλές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, όπως είπαν πολλοί ομιλητές. Μπορούμε να μειώσουμε τα ανώτατα όρια, που είναι μια απότομη και βίαιη λύση, ή μπορούμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και να ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουν οι δυνάμεις του ανταγωνισμού και μακροπρόθεσμα θα ρυθμίσουν την αγορά. Η δική μας ένωση, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, η BEREC, πάντοτε ακολουθεί μια συνετή προσέγγιση. Αναλύουμε τα στοιχεία και παραμένουμε σε μια φρόνιμη προσέγγιση. Δεν λέμε ότι δεν θα γίνουν όλα αυτά. Θα γίνουν για τους επιχειρηματίες και για αυτούς που συχνά χρησιμοποιούν την περιαγωγή. Μπορούν μέσω του ανταγωνισμού να επιτύχουν κάποιες καλύτερες τιμές, αλλά ο μεγάλος αριθμός των καταναλωτών στην αγορά δεν ξέρω πόσο θα επωφεληθούν. Αν δηλαδή ο ανταγωνισμός μεσοπρόθεσμα θα ωφελήσει και τους απλούς καταναλωτές. Οπότε το δίλημα κάπου εκεί κινείται και κατά συνέπεια ο Μπέρεκ θεωρεί ότι τα ανώτατα όρια που πρότεινε η Επιτροπή μάλλον είναι πολύ γενναιόδωρα. Δεν προστατεύουν επαρκώς τους καταναλωτές από το ενδεχόμενο να μην εμφανιστούν οι συνέπειες του ανταγωνισμού στην αγορά σύντομα. Και γι' αυτό ο Μπέρεκ ε, κάνει μια έκκληση να μειωθούν τα ανώτατα όρια που πρότεινε η Επιτροπή. Κάποια άλλα σημεία που έχω σημειώσει τώρα από τη συζήτηση. Αναφέρθηκε το πρόβλημα που θα το αποκαλέσω πρόβλημα Apple και Google. Είναι μάλλον νομικό το πρόβλημα και δεν είναι θέμα που μπορεί ένας τεχνοκράτης να σχολιάσει αν το θεωρεί καλό ή όχι. Η τεχνοκρατική ανάλυση είναι ότι οι μεγάλοι παίκτες από όπου και αν έρχονται, αν μπουν στην αγορά και ασκήσουν πίεση στον ανταγωνισμό, θα ωφελήσουν τελικά τους καταναλωτές. Αυτό είναι η δική μου γωνία. Τέλος, για την ε, απαλλαγή, για αυτή την πρόταση ε, για τις εταιρείες που είναι πρόθυμες να προσφέρουν μία τιμή όπου η τιμή περιαγωγής θα είναι κάπου κοντά και μπορούμε να το συζητήσουμε τι σημαίνει κοντά αλλά αν είναι έτοιμες οι εταιρείε, αν είναι πρόθυμες να προσφέρουν τιμές κοντά στις εγχώριες τιμές, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποδεσμοποίησης. Ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ ισχυρό και επιτυγχάνει νομίζω αυτό το οποίο όλοι επιθυμούμε. Τιμές περιαγωγής να είναι κοντά στι εγχώριε τιμέ, ώστε να μην, μπορούν να, ανησυχούν, να μην ανησυχούν οι καταναλωτέ και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά του τηλέφωνα όταν βρίσκονται στο εξωτερικό σε περιαγωγή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιε συνέπειε. δηλαδή αυτό θα λειτουργήσει πολύ πιο εύκολα σε χώρε όπου οι εγχώριε τιμέ είναι υψηλέ, και όχι σε χώρε όπου οι εγχώριε τιμές είναι χαμηλέ. Και το κόστος χονδρικής η τιμή χονδρικής της περιαγωγής μάλλον είναι πολύ υψηλή, υψηλότερη από την εγχώρια τιμή. Υπάρχουν χώρες όπου το περιθώριο λοιπόν μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν είναι μεγαλύτερο και μπορούν πιο εύκολο να το κάνουν και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για να σας δείξω πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές στην Ευρώπη. Ο Μπέρεκ πέρυσι έκανε υπολογισμού και η χώρα με τις υψηλότερες τιμές για φωνητικές υπηρεσίες ε, Τε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, τελειώνω μέση τιμή 17 λεπτά του ευρώ το λεπτό και η χαμηλότερη χώρα 2 λεπτά του ευρώ το, αναλεπτό ομιλίας. Επομένως, σε μια χώρα όπου οι τιμές είναι 17 cents, 17 λεπτά, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από ό,τι στις χώρες όπου είναι 2 cents το λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε την ακρόαση μέσα σε κάποιο χρονικό περιθώριο. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κορόλα και στην κυρία Νίμπλιο στη συνέχεια για να κλείσουν τη συζήτηση. Παρακαλώ. Uh, <clears throat> ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχουμε κάνει και με τις κατευθυντήριες γραμμές στην Επιτροπή Μικό. Αν δούμε το σημερινό αντίκτυπο του σημερινού αντίκτυπου βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η τιμή και για τις κλήσεις και για τα SMS περιεγωγής. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ε, λιανικής ε, βρίσκονται κοντά στι μέγιστε τιμέ και δεν υπάρχει ανταγωνισμός η Κομισιόν στους στόχους της για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο έχει αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ περιεγωγής και των εθνικών ε, τιμών θα πρέπει να φτάσει στο 0, κοντά στο 0 μέχρι το 2015. Για να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο αυτό είναι απαραίτητο να βρούμε μια λύση που να εγγυάται τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς περιεγωγής ε, και μετά από αυτή την ημερομηνία τα διαφορετικά μέτρα και τα νότα τα όρια τιμής δεν μπορούμε να τα ε, δούμε ξεχωριστά και το ίδιο ισχύει για τα ανώτατα όρια στη χοντρική και στη λιανική. Αν θέλουμε μια διερθωτική λύση που θα φέρει ανταγωνισμό, θα πρέπει να αφήσουμε επαρκές περιθώριο μεταξύ των τιμών χοντρική και λιανικής ε, για να προσελκύσουμε νέους παίκτες στην αγορά έτσι ώστε οι τιμές ε, να είναι λογικές ε, ως προς το κέρδος και να μπορούμε να άρουμε τα ανώτατα όρια αν αντίθετα αποφασίσουμε μέσω τη νομοθεσία, να ρυθμίσουμε τιμέ και μέσω τη νομοθεσία, να τι φέρουμε κοντά στι εθνικέ τιμέ μπορούμε ε, να ξεχάσουμε την αγορά και επίση θα πρέπει να σεβόμαστε την νομοθεσία τιμών στο μέλλον. συζητούμε τις διάφορες διορθωτικές ε, λύσεις, ε, όλες ε, αυτές που παρουσιάστηκαν οι λύσεις, όπως το local breakout και άλλες λύσεις, έχουν πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και μειονεκτήματα. Πρέπει να δούμε όμως ποια θα λειτουργήσει καλύτερα μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν θα ήταν γελίο να καθορίσουμε ποια νομοθεσία και ποια τεχνική λύση θα πρέπει να επιλέξουμε γιατί μπορεί να καταλήξουμε στο να δημιουργούμε νομοθεσία που, θα ήδη, που ήδη θα είναι ξεπερασμένη τη στιγμή της εφαρμογής. Η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και έτσι λοιπόν στην νομοθεσία μου ΙΜΚΟ εγώ αποφάσισα την τροποποίηση του κανονισμού αναφέροντας απλώς τα ουσιαστικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει τελική λύση όπως έκανε και η κυρία Νίμπλερ για το θέμα αυτό νομίζω ότι πρέπει να, να συνεχίσουμε να έχουμε θέμα τιμών λίγα χρόνια μετά το 2016 γιατί θα χρειαστεί χρόνος για να εξελιχθεί η αγορά. Για την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια. Η διαφάνεια των τιμών ε, έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους κανονισμούς περιεγωγής, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η πρόοδος αυτή οι καταναλωτέ, ε, θα πρέπει να εγγυόμαστε παροχή πληροφοριών στους καταναλωτέ με έναν ε, ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, να μπορούν οι καταναλωτέ εύκολα να συγκρίνουν ε, τι τιμέ και να μπορούν να αλλάζουν παρόχους των υπηρεσιών roaming, εγώ πρότεινα ε, ένα ανώτατο όριο τιμής ασφαλείας 50 ευρώ ή ένα ε, προσωποποιημένο για να αποφευθούν ε, δυσάρεστες εκπλήξεις θα πρέπει να επεκταθεί και στην περιαγωγή. Επίσης ο καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνει μια κοινοποίηση από τον πάροχο όταν πλησιάζει το ανώτατο όριο ε, της περιαγωγής. Επίσης, έχω προτείνει επιτεταμένα μέτρα για ε, τους προπληρωμένους ε, γιατί πολλές φορές ακόμη και με τέτοια συμβάσεις ε, μπορεί κάποιος ε, να έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Και θέλω να πω ότι η ενημέρωση του καταναλωτή αντικατοπτρίζεται σωστά στην πρόταση της Κομισιόν, όμως ε, θα έπρεπε με αυτή την διατύπωση να έχουμε δράξει την ευκαιρία να πετύχουμε μια σαφέστερη διάρθρωση του κανονισμού για την ενοποίηση όλων των διατάξεων ε, για την προστασία των καταναλωτών και για τις άρθρες εκπλήξης τους ε, λογαριασμούς και επίσης και για τις απαιτήσεις διαφάνειας που εφαρμόζονται σε όλες τις που ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στην Αγγέλικα ε, Νίβλε από την Επιτροπή Ήτρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, να δούμε πώς μπορούμε κατά το βέλτιστο τρόπο να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο από την Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών, την ΜΠΕΡΕΚ. Θα μείνουμε σε επαφή γιατί νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για όλες τις παρεμβάσεις σας. Ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμες από όλους τους τομείς που προέρχονταν και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή λύση που θα ενισχύει τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη και θα προσφέρουμε λογικές τιμές στον καταναλωτή ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη με λογικές τιμές. Ευχαριστώ πολύ την Αγγέλικα Νίμπλερ και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον Μάρκομ Χάμπορ, πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χέρμπερτ. Είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την Επιτροπή μου ε, που μας καλέσατε να πούμε και τη δική μας άποψη από την πλευρά των δικαιωμάτων των καταναλωτών ε, και των χρηστών και την προστασία των καταναλωτών. Βλέπω και την Πιλάρ Καστίγιο. χαίρομαι πολύ γιατί μαζί είχαμε εξετάσει τη δέσμη μέτρων για τα τελεπικοινωνιακά. Κάποιε καταληκτικέ παρατηρήσει. Ε, δεν ήμουν εδώ σε όλη την ακρόαση, αλλά ήμουν πρόεδρο σε αστυνομική επιτροπή όπου είχαμε και την παρουσία τη Πολωνική Προεδρία. Μια πιο γενική παρατήρηση για να ξεκινήσω. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό ε, που συμμετέχει και η Μπέρεκ ε, σε, αυτή την, αυτού του φακέλου. Από τότε που συγκροτήθηκε αυτός ο οργανισμός θεωρήσαμε ότι όλοι οι εθνική. Ε, ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά ε, στην ε, διαδικασία χάραξης πολιτικής. Αυτό θα είναι καλό για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, για τι αγορέ. Έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τον κύριο που είναι εδώ και τώρα και στους προηγούμενους δύο γύρους του κανονισμού για, τον, για την περιαγωγή. Τότε ήταν στην αντιπροσωπεία του Βασιλείου, βέβαια. Τώρα, εξακολουθεί η Μπέρεκ να μαζεύει δεδομένα για το κόστος. Και οι δύο ε, αυτό που θέλουν είναι να έχει πλήρη πρόσβαση στη, στα στοιχεία αυτά και στο μέλλον η, ε, η Μπέρεκ για να μπορεί να εκτελεί σωστά το έργο της. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά πάνω στη, στα δικαιώματα των χρηστών και θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν σαφή, έγκαιρα και εύληπτα στοιχεία για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, αν μπορούν να επιλέξουν πάροχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Κόρχαλα και νομίζω και η κυρία Νίμπλερ το έθεσαν και το έχουν περιλάβει και στις εκθέσεις τους. Αυτό είναι σημαντικό. Η δεύτερη παρατήρηση από τη δική μας πλευρά συνδέεται και με το έργο που έχουμε επιτελέσει και στο παρελθόν μαζί, είναι ότι έχουμε ασκήσει πολλή πίεση για τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν ε, οι καταναλωτέ να αλλάζουν πάροχο. Μια από τι λύσει που έχει τεθεί εδώ επιτάπητο είναι οι καταναλωτέ να μπορούν να επιλέγουν ξεχωριστό πάροχο που θα παρέχει τι υπηρεσίε περιαγωγή. Και θα πρέπει να είναι απολύτω σαφέ και σίγουρο ότι αυτή η δυνατότητα αλλαγής παρόχου ε, να μπορεί να γίνει τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Η Ρίτα νομίζω προτείνει κάποιο πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα, κάποια πιο σύντομη προθεσμία. Αυτό μπορούμε να το αφήσουμε βέβαια κατά μέρο προς το παρόν, γιατί θέλουμε να μας πει η Μπέρεκ ποιες είναι οι τεχνικές προϋποθέσεις, τεχνικοί όροι. Όταν είχαμε ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή μα μεταξύ άλλων είχε τονίσει ότι θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ε, η αλλαγή ε, παρόχου, η φορητότητα δηλαδή, να γίνεται με πολύ πιο γρήγορο τρόπο η όλη διαδικασία. Και υπήρξε σημαντική βελτίωση. Μέσα σε 24 ώρες μπορεί κανείς ε, τώρα να αλλάξει πάροχο. Άρα θα πρέπει η δυνατότητα επιλογής παρόχου να συνοδεύεται με ταχεία και εύκολη αλλαγή χωρίς καθυστερήσεις ώστε η εναλλακτική προσφορά να μπορεί να παρέχεται χωρίς περιορισμούς ή μειονεκτήματα για τον καταναλωτή. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που θέλουμε να το επεξεργαστούμε. Δεν θέλω να επισέλθω στη συζήτηση ε, σε ό,τι αφορά τις ανώτατες τιμές. Να πω όμως ότι κατ' εμέ είναι σημαντικό το καθεστώς με τις ανώτατες τιμές να παραμείνει σε ισχύ όσο χρειάζεται για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Σίγουρα οι πλευρές οι δύο στις οποίες ανήκουμε διαφωνούν σε κάποια πράγματα, αλλά Νομίζω ότι η Επιτροπή μας, βλέποντας και την έκθεση της κυρίας Κόρχολα, είναι υπέρ μιας λύσης που θα επιτρέψει επαρκή περιθώρια για να μπορούν να γίνουν νέες επενδύσεις και να βρεθούν νέες λύσεις. Επίσης είμαστε υπέρ της θέσης της υπηρεσία Μπέρεκ που λέει ότι δεν έχει γίνει επαρκής ανάλυση για κάποιες τις λύσεις ακόμη και δεν είναι χρόνος ε, τώρα να βιαστούμε ε, με μη δοκιμασμένες λύσεις, αν δεν έχουμε τεκμηρίωση, αν δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό να εξακολουθήσει να ισχύει αυτό το καθεστώς αυτών των όριων. Και ολοκληρώνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Μια λύση που δεν θα απαιτεί ακόμα μια σειρά κανονισμών ε, για την περίοδο 4, 5, 6 και θα έρχεται εδώ εκπρόσωπος της Μπέρεκ μέχρι να πάρει σύνταξη για να μας ε, λέει ε, για μια ακόμη για αυτά τα περιθώρια. Όχι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν έχουμε εξοπλιστεί, δεν ε, έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να μπορεί να λειτουργεί αγορά και να είναι καινοτόμα και να παρέχει στο μέλλον νέε λύσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει για να μπορέσουν να επιτευχθούν όλα αυτά, να του δώσουμε εμείς τη δυνατότητα, την ευκαιρία. Και ευρύτερα να δούμε και τι θα γίνει και στην εγχώρια αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Ξεκολουθούμε να έχουμε σε πολλές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τις τιμές με πολλούς παρόχους. Μιλάω για τη λιανική τιμή. Μόνιμη δηλαδή ρύθμιση τη κινητή τηλεφωνία. Πρέπει να βρούμε κάποια λύση. και αυτή η ιστορία εδώ με τους νέους παρόχους, να έχουμε ένα καθεστώς ώστε να μπορούν να υπάρχουν και αυτοί οι εικονικοί πάροχοι ε, για το roaming. Αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και την και την τηλεφωνία και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Προσβλέπω λοιπόν ε, στην συνέχιση του έργου και της συνεργασίας μας ε, και σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσετε δική μας επιτροπή. Να ευχαριστήσω και για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που άκουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Μάλκολμ, ευχαριστούμε όλους για τις παρεμβάσεις σας και για την εξαιρετική συνεργασία. Χαιρόμαστε για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να κλείσουμε την ακρόαση. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και πάλι. χωρίς να χρειάζεται να ξανανοίξουμε τις συζητήσεις ε, που έγιναν ε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Αύριο είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών στις 12, 12 και κάτι. 12 η ώρα λοιπόν η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών γιατί θα πρέπει η γραμματεία να έχει το χρόνο για να μπορέσουμε τον Ιανουάριο να καταλήξουμε κάπου. Δεν γίνεται διαφορετικά γιατί θέλουμε να καταλήξουμε σύντομα σε κάποια λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κλείνει λοιπόν και το σημείο 12 της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της άλλης επιτροπής και τους προσκεκλημένους μας και τις εισηγήτριες. Και στην επιτροπή μας περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Äh, Το επόμενο σημείο της μείσης διάταξης είναι η συζήτηση με την Πολωνική Προεδρία που όμως δεν έχει ακόμη γιατί εμείς καταφέραμε και τελειώσαμε νωρίς. Ähm, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί δεν έχει έρθει ο Πολωνός εκπρόσωπος. Μικρό διαλυματάκι λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Στις και μισή. Όχι στις και μισή. Έξι παρατέταρτο το έχουμε προβλέψει. Έξι παρατέταρτο λοιπόν. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν ξαναγυρίσετε. Μην με αφήσετε μόνο με την Πολωνική Προεδρία. Ε, ξέρετε, καμιά φορά και εγώ το κάνω και φεύγω, αλλά μια και είσαστε εδώ, να υποφεληθώ και να σας το πω. Ας ξανάρθει κάποιος, όποιος μπορεί και βουλευτές και βοηθοί. Not laughing too much. Okay. Θα κάνω συνεδρίαση με τους διερμηνείς. Διερμηνείς είναι περισσότεροι από τον πρόεδρο. Δύο, δύο βουλευτές και 60 διερμηνείς. Κερδίζουν οι διερμηνείς. Θα ήθελα, μια και είμαι εδώ, να σα ευχαριστήσω τα δυόμιση χρόνια που είμαι εδώ πρόεδρος, γιατί πάντοτε χαίρομαι που σας ακούω. Πάντοτε πάνε όλα πολύ καλά με τη διερμηνία. Σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Κάθε ευτυχία στην καινούργια χρονιά και καλή συνέχεια των εργασιών μας ε, εδώ. Ευχαριστούμε και οι διερμηνείς στον Πρόεδρο. Ξέρω ότι εγώ συνήθως μιλάω γρήγορα, εκτός από αυτό το σημείο τριβής, κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν σας ταλαιπωρώ. Πάντως από ό,τι ξέρω οι διερμηνείς για μένα λένε ότι μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε όλοι μαζί την Πολωνική Προεδρία. Είμαστε εδώ ο κύριος Σοντή και εγώ και περιμένουμε την Πολωνική Προεδρία. Okay. Das war's. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω ότι θα έρθουν και άλλοι κατά τη διάρκεια των συζητησιών μας. Αλλά σήμερα, όπως είπα ήδη στην ε, κυρία Υφυπουργό, είχαμε διάφορες συνεδριάσεις παράλληλες ώρες και πολλοί συναδέλφοι σίγουρα κολλείονται και δεν μπορούν να είναι παρόντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μαγδελένα Πά και χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σχετικά με την Πολωνική Προεδρία στα θέματα που αφορούν τη δική σας αρμοδιότητα. Σα δίνω το λόγο λοιπόν για να ξεκινήσετε εσεί και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά. E, e, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μου δίνετε η δυνατότητα ε, να ε, είμαι σήμερα στην Επιτροπή σας για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας τα θέματα τηλεπικοινωνίας ε, και ε, ψηφιακής διαχείρισης. Ολοκληρώνεται τώρα το εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας. Αυτό το εξάμεινο δεν ήταν το πρώτο εξάμεινο με οικονομική κρίση στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η κατάσταση ε, γύρω μας και γι' αυτό πρέπει να αντιδρούμε όχι μόνο γρήγορα αλλά και με καινοτομία. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της προσέγγισής μας. Στη σύντομη παρέμβασή μου θα μιλήσω όχι μόνο για τη δική μας συνεργασία, αλλά θέλω να αναγνωρίσω και τη δική σας δέσμευση και συνεισφορά και θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία μας. Τα καταφέραμε μαζί. Εσείς και εμείς, η Πολωνική Προεδρία, από κοινού νομίζω ότι επιτύχαμε να, έχουμε το πρώτο να εγκριθεί το πρώτο πρόγραμμα RSPP και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντική η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει. Το πιο σημαντικό αντικείμενο της Προεδρίας μας ήταν η ταχεία έγκριση του πρώτου προγράμματος για το ραδιοφάσμα. Μία συμβιβαστική λύση για αυτό το δύσκολο θέμα ε, σημαίνει την απελευθέρωση τεράστιου δυναμικού, κυρίως για το ραδιοφάσμα, για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά λέγει ότι ο τομέας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ένας τομέας που μπορεί να συνεισφέρει πολύ στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό ήταν μεγάλο επίτευγμα το να εγκριθεί γρήγορα το πρώτο πρόγραμμα RSPP. Σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το έγγραφο για το RSVP. Χρειάστηκε πολλή δουλειά από εμπειρογνώμονες σε ομάδες εργασίας. Έγιναν και πολλές τεχνικές συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Έγιναν ε, πολλές διαπραγματεύσεις και με τον Πρόεδρο κ. Ρόιλ και με τον ε, κ. Χόκμαρκ και τελικά τα καταφέραμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας για αυτό το πρόγραμμα RSPP. Είναι σημαντική η συνεισφορά μας για τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανταγωνιστικότητα και για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ως Προεδρία ασχοληθήκαμε και με την περιαγωγή, με την καθολική υπηρεσία και με, τη, με το δεύτερο δίκτυο, με την ουδετερότητα του δικτύου και με το μέλλον του ΕΝΙΖΑ. Όσον αφορά την περιαγωγή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πρέπει να πω ότι ήταν μία από τις βασικές μας προτεραιότητες και για μας είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών αφενός ε, που τους ενδιαφέρει η περιαγωγή, γιατί οι καταναλωτές θέλουν να υποφεληθούν από τις υπηρεσίες περιαγωγής και από την άλλη πλευρά ε, ε, βρίσκονται οι πάροχοι δικτύου που και αυτοί έχουν τα συμφέροντά τους. Ήταν σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον κανονισμό που θα μειώσει τα τέλη για τους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική αγορά και σε αυτό συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς που θα πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές και θα δίνουν στις εταιρείες κίνητρα για καινοτομία. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. Στην ομάδα εργασίας τα κράτη-μέλη συμφωνούσαν όσον αφορά το νέο σχέδιο κανονισμού. Και στην τελευταία συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου η πλειοψηφία των Υπουργών δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να δώσουν την εντολή στις διοικήσεις τους να προωθήσουν και να υλοποιήσουν αυτό τον κανονισμό το ταχύτερο δυνατόν. υπάρχουν ε, τα θέματα των διαρθρωτικών λύσεων ε, πάνω στα οποία δουλεύουν οι τεχνικές επιτροπές σε τεχνικό επίπεδο ε, για να υλοποιήσουμε την αποδεσμοποίηση και τα κράτη-μέλη δουλεύουν πάνω στο θέμα της αποδεσμοποίησης και θα ακολουθήσουν αργότερα οι τεχνικές λεπτομέρειες. Κλείσαμε το θέμα της περιαγωγής με μια έκθεση προόδου η οποία εγκρίθηκε στις 13 Δοδεκάτου και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία την οποία είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι σήμερα οργανώσατε και μια κρόαση με βάση την έκθεση της κυρίας Νίμπλε και ελπίζω ότι στην αρχή του επόμενου έτους, κατά την Δανική Προεδρία, θα καταλήξουμε σε συμφωνία και ο, επόμενο, ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2012. Ως ε, υπουργό για τις τηλεπικοινωνίες σας εγγυώμαι ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξη της Πολωνίας και τη συνεργασία μας ε, ε, στα θέματα αυτά. Ελπίζω ότι το συντομότερο δυνατόν θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους καταναλωτές ε, και όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εποχές οικονομικής κρίσης όπως η τωρινή είναι σημαντική η περαιτέρω πρόοδος της ψηφιακής αγοράς. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια δικτύου και την ασφάλεια των πληροφοριών και αυτή ήταν άλλη μία πρωτοβουλία μας ενίσχυση και εξυγχρονισμός του ΕΝΙΖΑ. Συνεργαστήκαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη. Ε, και δεν έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις τις οποίες έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη. Τα νέα καθήκοντα του ΕΝΙΣΑ συμπεριλαμβάνουν τη συνεργασία με το ΣΕΤ και τα ΣΥΡΤ για να προωθήσουμε την ασφάλεια δικτύων. Ε, στον ΕΝΗΣΑ συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και υποστηρίζουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι καλά και περιμένουμε ε, την ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε που έχει προγραμματιστεί για το Μάρτιο του 2012. Ελπίζω ότι η Δανέζικη Προεδρία θα μπορέσει να ολοκληρώσει τότε το θέμα. Η Πολωνική Προεδρία διεξήγαγε μια συζήτηση και για το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας. Ήταν ένα από τα θέματα του τρίο της Πολωνικής, Δανέζικης και Κυπριακής Προεδρίας. Και στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία και να παρέχουμε εγγύσεις για τα δικαιώματα των χρηστών. Ακούσαμε τις απόψεις της Επιτροπής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση στις 23 Νοεμβρίου για την Καθολική Υπηρεσία και παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχει κάποια βασική ανάγκη για κάποια τροποποίηση, έχει προγραμματίσει την δημοσιοποίηση ενός εγγράφου για την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο με εγγύησεις ε, για την ε, ορθή παροχή ε, υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ισορροπημένη προσέγγιση. Χρειαζόμαστε επενδύσεις κυρίως στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. και Παράλληλα, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε υπερβολικά πολλές υποχρεώσεις στους παρόχους. Όσον αφορά την ουδετερότητα δικτύου, υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση της Επιτροπής και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με την ανακοίνωσή της αυτή, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα κατάλληλα δεδομένα που θα ανακοινώνονται και από την ε, Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών, από την ε, Μπέρεκ. Με βάση την ε, εξέταση αυτών των στοιχείων θα εξετάσει περαιτέρω η Επιτροπή τα θέματα ουδετερότητας δικτύου. Η Πολωνική Προεδρία στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου αναγράφεται σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση της Επιτροπής. Και σε αυτό το έγγραφο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τονίζεται η σημασία του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου, ούτω ώστε να παραμείνει το διαδίκτυο κάτι το ισχυρό και αξιόπιστο με προστασία των βασικών ελευθεριών, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του επιχειρήν. Ως Προεδρία χαιρετίζουμε και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ουδετερότητα του δικτύου και υπάρχει το ψήφισμα από τις 17 Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό είναι αρκούντος θετικό προς την ανακοίνωση της Επιτροπής. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας των πληροφοριών έλαβαν χώρα διάφορες εκδηλώσεις στην Πολωνία και θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε αυτές. Στις 19 και 20 Οκτωβρίου οργανώσαμε μια συνάντηση υπουργών για τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Συμμετέσχουν υπουργοί τηλεπικοινωνιών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι των διεθνών οργανώσεων και συνδέσμων τηλεπικοινωνιών, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες και άλλοι. Στόχος ήταν η παρουσίαση των μελλοντικών εξελίξεων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλήσαμε για το ραδιοφάσμα με βάση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για το συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και παράλληλα τονίσαμε τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ηλεκτρονική επικοινωνία και τα δίκτυα νέας γενιάς, τα NGA. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γκίναρ Χέκμαρκ για τα σχόλιά του και για την πολύ ζωντανή παρέμβαση που έκανε κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου αυτού. Η συνεδρίαση αυτή ολοκληρώθηκε με μια διακήρυξη σχετικά με το διαδίκτυο. Προσυπέγραψαν πολλοί από τους ε, παρευρισκομένους και θα συνεχίσει η συγκέντρωση υπογραφών ε, για την ε, διακήρυξη αυτή. Είναι μια πολύ σημαντική διακήρυξη και προετοιμάζεται και μια διάσκεψη στη Γενέβη, η Διεθνής Διάσκεψη Ραδιοφάσματος, που θα πρέπει κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια να προσδιορίζει τις βασικές γραμμές. Υπεγράφει λοιπόν αυτή η διακήρυξη και από τα κράτη-μέλη και από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελέσει αυτή η διακήρυξη μια καλή βάση για την πρόθεση των εργασιών που θα ξεκινήσουν στη Γενέβη το 2012. Η Πολωνία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε την έκτη Υπουργική Διάσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για τις διαμεθοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στόχος μας ήταν η συγκέντρωση όλων των εμπειριών των κρατών μελών και η ενασχόλησή μας με τις προκλήσεις που τίθενται για την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Υπάρχει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τέθησαν στόχοι για το 2011 έως 2015. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στρέφονται γύρω από αυτό το θέμα και στη διάσκεψη συζητήσαμε τα ωφέλη που θα μπορούσαν να υπάρξουν για τους πολίτες και για τους καταναλωτές καθώς και για τις επιχειρήσεις και αναφέρθηκαν και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παράλληλα με αυτή τη διάσκεψη διεξήχθη και μία συνάντηση υπουργών για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, έκθεση των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών έργων που προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ήταν μεγάλη η απήχηση αυτής της διάσκεψης. Συμμετείχαν περίπου 800 εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εθνικές και περιφερειακές οργανώσεις, από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Παγκόσμια Τράπεζα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, εκπρόσωποι από τον τομέα της εκπαίδευσης, από τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το Υπουργείο μας προετοιμάζει τα λεπτομερή πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα βάλουμε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στο διαδίκτυο. οι δραστηριότητε μας κάλυψαν και διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέσχομαι το Σεπτέμβριο σε μια διάσκεψη στο Ναϊρόμπι. Είχε προετοιμάσει η Προεδρία ένα έγγραφο της Προεδρίας, το οποίο είχε προετοιμαστεί από τα κράτη-μέλη. Μεταξύ άλλων, τονίστηκαν τα ενδιαφέροντα πολλών φορέων όσον αφορά την ελευθερία στο διαδίκτυο και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ε, με άλλες χώρες και με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και τώρα η επόμενη Προεδρία θα είναι η Δανέζικη Προεδρία που την περιμένουν πολλές προκλήσεις. Ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε και την επόμενη Προεδρία όσο υποστηρίξατε εμάς και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ganz Σας ευχαριστούμε πολύ λεπτομερέστατη η παρέμβασή σας και σας ευχαριστούμε και εμείς για την πολύ καλή συνεργασία μας. Ήταν ε, μια περίοδος με πολύ σημαντικά πολιτικά προγράμματα. Ε, μερικές φορές ήταν πιο εύκολο, άλλες φορές ήταν πιο δύσκολη η κατάσταση. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο Όντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Να σας πω καταρχήν ε, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η σοφία του πολωνικού λαού σας ε, ανέθεσε την εξουσία στη χώρα σας γιατί ήταν καταπληκτική η προεδρία σας και σήμερα κάνουμε την αποτίμηση και νομίζω ότι η κυβέρνησή σας μπορεί να είναι πολύ περήφανη για το έκανε στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για το χαρτοφυλακείο Εγώ θέλω να σας εκφράσω μια ανησυχία που αισθάνομαι ότι στο βαθμό που οι επιστημονικές ιδιοφυΐες μας παρουσιάζουν νέες τεχνολογίες, οι πολίτες έχουν το συνέστημα ότι ο ψηφιακός κατακαιρματισμός δεν επιλύεται ποτέ. Και υπάρχει αυτό το αίσθημα δηλαδή ότι δεν υπάρχει μεταχείριση των πολιτών, ε, δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες οπουδήποτε καν βρίσκουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και εμείς, πολιτική εξουσία, θα πρέπει να βρούμε τα πολιτικά και τα χρηματοοικονομικά μέσα για να δώσουμε αυτή την ε, διαβεβαίωση στους πολίτες. Ε, σήμερα το απόγευμα συζητήσαμε πολύ για ε, τις τιμές, για τα τέλη της περιαγωγής ε, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια κίνηση για να μειωθούν οι τιμές των παρόχων, όμως ξεχνάμε από την άλλη ότι οι συμπολίτε μα θα ήθελαν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι οι επενδύσει γίνονται για να μπορούν να έχουν αυτή πρόσβαση στι υπηρεσίε. Γιατί αν δεν επιλύσουμε το πρόβλημα τη πρόσβαση ε, στι ψηφιακέ υπηρεσίε, τότε ο πληθυσμός ε, θα συνεχίζει ε, να κατακλείζει τα αστικά κέντρα με όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε, ασφάλεια, εκπαίδευση κτλ. Και μετά από αυτούς τους 6 μήνες ε, προεδρίας, θέλω να πω, η πολιτική της Επιτροπής και των κρατών μελών. Σέβεται αυτή την αναγκαιότητα του συνόλου της χορταξίας ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επικράτειας με την παροχή ευκαιριών και εδώ έχουμε μια συνέπεια. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσουμε την αγορά Πρέπει να οργανώσουμε τις αγορές. και οι κυβερνήσει των κρατών μελών ε, καθορίζουν τι υποχρεώσεις τη κάλυψη. Πώ ε, λοιπόν θα ρυθμίσουμε αυτή την ασυνέπεια αν μειώσουμε τα τέλη για να ικανοποιήσουμε τον καταναλωτή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή για το περιαγωγή και αφαιρούμε από την άλλη εισόδημα από τους παρόχους και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις κυβερνήσεις ε, για τις υποχρεώσεις κάλυψης και εθνικές κυβερνήσεις, ε, τουλάχιστον αυτή είναι η περίπτωση της δικής μου χώρας. Στο πρόσφατο παρελθόν ε, έλεγε θα καλύψετε το 80% του πληθυσμού, σε προθεσμία σε χρονοδιάγραμμα 100. Όμω αυτό δεν είναι ε, αποδεκτό, γιατί αν ζείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται και όπου μένω εγώ παραδείγματο χάρη, στο ψήφο του Μπουλβά, ε, δεν έχετε ίσες ευκαιρίε και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου πείτε τι πιστεύετε γι' αυτό και θέλω να σας θέσω και μια ερώτηση για την Τρόικα, Πολωνία, για το τρίο των Προεδριών, Πολωνία, Δανία, Κύπρος, αλλά εσείς απαντήσατε για ε, απαντώντα στο ε, θέμα των καθολικών υπηρεσιών, τη καθολική υπηρεσία. Και πάλι θέλω να σα ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά τη κυβέρνησή σα, αλλά και το εκεί εξαιρετικό έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκάι για να απαντήσει. Ε, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας ε, λόγια. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος της ε, κυβέρνησής μου. Ελπίζουμε ότι στη χώρα μου η κυβέρνηση μου θα συνεχίσει να έχει την εξουσία και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, γιατί κατά τέτοιο σε περίοδο κρίσης ε, εγγυάται τη συνέχεια γιατί δεν ε, υπάρχουν αλλαγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι λοιπόν ελπίζω τα επόμενα έτη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή σα σε σχέση με τις επενδύσεις για την πρόσβαση στα δίκτυα και σε σχέση με την αναγκαιότητα να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών μας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και ευρύ θέμα και αναφέρθηκα στο θέμα αυτό όταν ε, μίλησα για τις καθολικές υπηρεσίες. Είπα ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, η οποία είναι δύσκολη βέβαια, μεταξύ της επιβολής ε, περαιτέρω άχθους ε, στους επιχειρηματίες και αφενός και τις, προσδοκίες, τις προσδοκίες της Κομισιόν και των κυβερνήσεων για την αύξηση των επενδύσεων αφετέρου, γιατί οι επενδύσεις ε, σε πιο σύγχρονες υποδομές, οπτικές σύνες, ε, παραδείγματος χάρη, η δυνατότητα πρόσβασης σε βριζονικές υπηρεσίες είναι τεράστιες. Οι επενδύσεις αυτές είναι τεράστιες και πρέπει να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες μας και να τους βοηθήσουμε καταργώντας τα εμπόδια στις επενδύσεις. Και Φυσικά θα πρέπει να θυμούμαστε ότι έχουμε και περιοχές όπου είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει κάλυψη εκεί και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, με τη δημιουργία κινήτρων Έτσι λοιπόν, ε, στις περιπτώσεις ε, που μιλάμε για αυτές τις ε, ζώνες, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους επενδυτές να επενδύσουν περισσότερο σε αυτές τις περιοχές. Αυτό γίνεται στη Γαλλία, αλλά γίνεται και στην Πολωνία. Και ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών αλλά και των εθνικών δημοσίων πόρων ενεργοποιούνται και διοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να συναυθούν ΣΔΙΤ, συμπιάξεις δημοσιοδιωτικού τομέα. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να έχουμε επενδύσει για να εγγυηθούμε την πρόσβαση των πολιτών στα πιο καινοτόμα δίκτυα, γιατί αυτή είναι η βάση. Ακόμη και αν ζει κάποιο σε μια πιο απομονωμένη περιοχή της Γαλλίας ή της Πολωνίας, είναι σημαντικό ο πολίτης ε, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, να μπορεί να, χάρη, να πάρει τηλέφωνο το γιατρό. Και για το τρίο των δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Εμείς ε, είχαμε μία συζήτηση για το μέλλον ε, της καθολικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ενός γεύματος των Υπουργών και η Προεδρία της Δανίας σίγουρα θα προωθήσει τις εργασίες αυτές Ε, σύμφωνα βέβαια και με τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις. Κυρία Χίμνα. Ναι, με ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την ε, κυρία Υπουργό, γιατί από ξέρω πρόσφατα να αναλάβατε αυτά τα καθήκοντα Εσείς ε, παρουσιάσατε διάφορες ε, πτυχές ε, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, μιλήσατε για τις επικοινωνίες, τις τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά έχω μια ερώτηση. Μια ερώτηση που συχνά μου θέτουν οι συμπολίτε μου. Δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε αυτή τη λεγόμενη ασφάλεια των δεδομένων. Ξέρουμε ότι σήμερα χρησιμοποιούν όλοι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις επικοινωνίες τους, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και για πληρωμές, για να παρέχουμε πληροφορίες, για να λάβουμε πληροφορίες. Έτσι λοιπόν γενικά οι πολίτες ανησυχούν κυρίως ε, για τις ε, τραπεζικές συναλλαγές Μία δεύτερη πτυχή που επίσης μάθησαν οι συμπολίτε είναι η ασφάλεια των ιατρικών πληροφοριών που στη συνέχεια ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για εκβιασμούς. Δηλαδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο αυτέ οι πληροφορίε. Ε, και πολλέ φορέ ε, δημιουργούνται τραγωδίες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξέρω αν υπό την Πολωνική Προεδρία ασχοληθήκατε ε, με το ζήτημα αυτό, αν το συζητήσατε κατά κάποιο τρόπο και αν θα, συνεχ... θα υπάρχει μια συνέχεια στο μέλλον. κατά τη διάρκεια αυτού του τρίου των προεδριών. Δηλαδή για να παρέχετε κάποιες εγγυήσεις, κάποια ασφάλεια στους πολίτες. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους πολίτες γιατί ξέρουμε ότι διαρροές ε, στο ίντερνετ ε, ε, αφορά και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και θέματα οικονομικής ασφάλειας. Πρόσφατα είχαμε κλοπές δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα. Ασχοληθήκατε λοιπόν καθόλου εσείς με το θέμα αυτό. Και αν όχι, έχετε κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά με το τι θα γίνει στο μέλλον, αν θα υπάρξει κάποια πρόταση σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Δεν το συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας γιατί αυτά είναι θέματα που άπτονται του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ε, πρέπει να ασχολούμεθα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας με αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το νέο πακέτο για τις ε, τηλεπικοινωνίες, ξέρω ότι είναι κάτι με το οποίο ε, ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με την υλοποίησή του και με, με τα θέματα ουδετερότητας δικτύου και ασφάλειας του διαδικτύου. και το νομικό πλαίσιο μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα ε, αδικήματα που μπορεί να είναι ε, του ποινικού δικαίου. Ε, στο νέο πακέτο νομίζω θα υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες, ιδίως για την ηλεκτρονική επικοινωνία. ο επιθεωρητής προστασίας δεδομένων και μια ειδική επιτροπή στην Πολωνία θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών και σε αυτά τα πλαίσια θα οργανώνονται και οι εργασίες για την ασφάλεια διαδικτύου. Εάν υπάρχουν ε, πληροφορίες, ε, λοιπόν διάθεση πληροφοριών σε άτομα που ε, δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοιες πληροφορίες, νομίζω ότι αυτά τα θέματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή. Εάν προκύψει κάτι τέτοιο, το επόμενο εξάμεινο που θα το εξετάζουμε και στην Προεδρία, θα αναθέσουμε τις αρμοδιότητες γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν, θα πρέπει να χειριστούμε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Först ber jag om ursäkt att jag inte lyssnade på genomgången. Jag blev förhindrad av en annan aktivitet. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, άκουσα το σύνολο της παρέμβασής σας, διότι είχα κάποιες άλλες αντλημένες υποχρεώσεις. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά από όσα άκουσα τουλάχιστον, πραγματικά ήταν πολλέ επιτυχίες επιτυχίε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την Προεδρία σα. Θα ήθελα να σα κάνω ένα ερώτημα πιο γενικού χαρακτήρα. Που έχει να κάνει και με τις δραστηριότητες ε, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τη έρευνα και της ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ο πολίτης και οι περιφέρειες τα διάφορα κράτη-μέλη ποια άλλη επίδραση θα έχουν. Στη Σουηδία εμείς, γιατί είμαι Σουηδός, έχουμε αναπτύξει την στρατηγική της Βαλτικής. Έχουμε λοιπόν κάποιες μορφές, ε, κάποιους τρόπους συνεργασίας ε, με τις περιφέρειες. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξή. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν του μουσιονομικού προγραμματισμού πώς θα προσπαθήσετε να βρείτε νέους μηχανισμούς. Γιατί προφανώς ε, το κονδύλιο στον προπολογισμό δεν μπορεί να αυξηθεί. Πώς θα έχουμε λοιπόν επαρκή αποτελέσματα για να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων συνεργασιών, περιφέρειες, ε, κράτη και πολίτες. Στην ε, Ευρώπη νομίζω ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Γι' αυτό και σας ερωτώ τι εμπειρίε υπάρχουν κατά την άποψή σα ήδη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία που θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε για να αναπτύξουμε νέα μοντέλα συνεργασίας ώστε οι ανταλλαγές μας να είναι πιο αποτελεσματικές στον τομέα τη δικό σας πεδίου αρμοδιοτήτων. Εφόσον επαναλαμβάνω, μέχρι το 2020 ο προπολογισμό μάλλον δεν μπορεί ε, να περιμένουμε ότι θα αυξηθεί. Τι συμπεράσματα λοιπόν, σε τι συμπεράσματα καταλήξατε και να σας ευχαριστήσω για μια κομφέρα για την εξαιρετική προεδρία σας. Ευχαριστούμε κύριε Γκάι, το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στην πρωτοβουλία των χωρών της Βαλτικής και η Πολωρία συμμετέχει Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και εκεί συναντούμαστε και συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα στο φόρουμ αυτό, αλλά αναρωτιέμαι πώς ακριβώς να απαντήσω στην ερώτησή σας, ε, γιατί εσείς είπατε ε, ότι πρέπει να δούμε αν έχουμε τους απαραίτητους ε, πόρους για να δημιουργήσουμε νέα βήματα συνεργασίας. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, Τίποτα δεν μπορεί να αντιποκατεστήσει μια άμεση επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Μια άμεση επαφή και μια καλή ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε αυτό και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και έτσι εργαστήκαμε. Οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο πάντοτε συνομιλούν με ανθρώπους που γνωρίζουν προσωπικά και με άτομα από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο. Και προσπαθούμε σχεδόν να γίνουμε φίλοι. Δηλαδή γίνονται απευθεία τηλεφωνήματα, ανταλλάσσουν πληροφορίε ε, και γνωρίζουν το άτομο και δεν ξέρουν απλώ το όνομά του και δεν ξέρουν σε ποιο πρόσωπο αντιστοιχεί. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και επειδή είναι καλέ σε διαπροσωπικές επαφές. Όμω αυτή είναι η αρχή στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σεμινάρια που οργανώνονται στις διάφορες ε, χώρες. Επίσης, πολλές φορές, ε, μπορώ να σας πω τους χάρη ότι το παρό, οργανώθηκε ένα σεμινάριο για ε, τις τηλεπικοινωνίες, για τις ε, σχετικές υποδομές των τηλεπικοινωνιών και κλήθηκαν και άτομα και από τα άλλα Κατόπιν, Είχαμε μια άλλη πρωτοβουλία για τις άμεσες επαφές όπου συμμετέχουν ε, και άλλα κρατή-μέλη όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και εκεί μιλάμε για τις συχνότητες και συζητούμε πώς ε, χρησιμοποιούμε, με το, πώς να χρησιμοποιούμε με το βέλτιστο τρόπο τις συχνότητες και σε ποια εναρμόνιση θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Επίσης έχουμε και ε, τον οργανισμό που είναι αρμόδιο για τις ε, τηλεπικοινωνίες και ο οποίος μας βοηθά στο να οργανώσουμε καλές πρωτοβουλίες σε διαπεριφερειακό επίπεδο και να προβούμε σε ένα διάλογο με τις άλλες χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν πάντοτε ανοιχτό πνεύμα και θέλουμε να συνεργαζόμαστε με όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε στην Επιτροπή μας, για τη συνεργασία μας μέχρι τώρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω τις ευχαριστίες όλων μας από την Επιτροπή μας να τις μεταφέρετε στην κυβέρνησή σας και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σε άλλους κύκλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστώ σε όλη την Επιτροπή και στους προσκεκλημένους και σε όλους τους συνεργάτες που συνεχίζουν να είναι ακόμη στην αίθουσα. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και πολύ καλή πρωτοχρονιά, καθώς και μια πολύ καλή επόμενη χρονιά, το 2012. Ελπίζω να είναι πολύ καλή χρονιά. Ίσως να έχουμε λίγο λιγότερη δουλειά εμείς, αλλά πάντοτε τα αποτελέσματά μας να είναι εξίσου ικανοποιητικά. Βλέπετε, οι πιο εργατικοί που έμειναν μέχρι το τέλος ακούνε και τι ευχαριστίες. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Εξ ονόματο της Πολωνικής Προεδρίας θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω, Πρόεδρε, και σας και όλου του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. θα ήθελα στα τέλη του 2012 να μπορούμε να ευχηθούμε κάτι εξίσου καλό για το 2013. Να είναι κάθε χρόνος εξίσου καλός με το προηγούμενο και ακόμη καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.